Λοιπόν, ξεκινούμε. Ψηφοφορίε. Πρώτα κανονισμού του Κοινοβουλίου είναι το πρώτο θέμα για ε, του τρόπου άσκηση του δικαιώματο και των πραγμάτων επιτροπή του Κοινοβουλίου. Ίσως ο κύριος Μάρτιν πριν αρχίσουμε να ψηφίζουμε μας ενημερώσει για την κατάσταση. Θα είμαι σύντομος, Πρόεδρε. Θα θυμάστε ότι στην Ολομέλεια τον Οκτώβριο του 2011 και με μεγάλη πλειοψηφία ζητήσαμε να αλλάξουν οι κανόνες των εξεταστικών επιτροπών για να παρασχεθούν δυνατότητες πρόσβασης στα δικαιώματα των εγγράφων, στο δικαίωμα να καλέσουμε μάρτυρες και να έχουμε καλύτερη εικόνα της έρευνας και της αληθοφάνειας των δεδομένων που εξετάζουμε. Η έκθεση αυτή ε, Πρόκειται μετά από μια εξεταστική επιτροπή που ανέδειξε ότι δεν μπορεί να φτάσει στην αλήθεια λόγω έλλειψης αυτών των εργαλείων. Είχαμε μια σειρά τριλόγων, ε, ο τελευταίος εκ ήταν πριν από ένα χρόνο και στο τέλος του τριλόγου ζητήσαμε από τις νομικές υπηρεσίες των τριών θεσμικών οργάνων να εξετάσουν το ενδεχόμενο μιας διατύπωσης δεκτής και στα τρία θεσμικά όργανα. Μετά από δέκα συναντήσεις των νομικών υπηρεσιών και μεγάλο αριθμό ανταλλαγή απόψεων, οι νομικές υπηρεσίες τη επιτροπή και του Συμβουλίου είναι φανερό ότι δεν έχουν πολιτική εντολή να διαπραγματευτούν τις αναγκαίες αλλαγές. Συστήνω λοιπόν να διαπιστώσουμε μέσω απόφαση σήμερα και στην Ολομέλεια ότι δεν θα ολοκληρωθεί η έκθεση αυτή μέσα στη θητεία του Κοινοβουλίου. Γιατί είμαστε ωστόσο το ψήφισμα και με τρόπο που θα μα επιτρέπει να διατηρήσουμε τα πλονεκτήματα και την πρόοδο που έχει ήδη επιτευχθεί και έγινε, επιτεύχθη πρόοδο στην πρόσβαση στα έγγραφα, στην χρησιμοποίηση των εγγράφων. Δεν θέλουμε να χαθούν αυτά. Η ιδέα είναι λοιπόν να διατηρηθεί ζωντανό το πνεύμα αυτού του στόχου για το επόμενο κοινοβούλιο που να διαπραγματευτεί από άλλη θέση ισχύω. Ωραία, προχωρούμε λοιπόν στην ψηφοφορία. Μία τροπολογία μόνο υπάρχει υπέρ. Κατά. Δύο. Τρεις. Αποχές. Μία αποχή. 22. υπέρ, 3 κατά, μία αποχή. Να προχωρήσουμε και στη δεύτερη ψηφοφορία για την πρόταση να καλέσουμε τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου να θέσει σε ψηφοφορία στη Σύνοδο του Απριλίου πλέον την πρόταση ψηφίσματος για την ε, τροποποίηση που αναφέραμε. Υπέρ, εν, ε, εν, υπάρχει αλλά καλύτερο είναι να το κάνουμε ούτως ή άλλως. Υπέρ, κατά, Τέσσερις κατά. Αποχές, κανείς. Ωραία. 22 έναντι 4. Προχωρούμε τώρα στην πρόταση τροποποίησης του κανονισμού του Κοινοβουλίου που τροποποιεί τα άρθρα 166 και 195 παράγραφος 3. Ο κ. Μέσσερ Σμιτ είναι εισηγητής. Ο κ. Μέσσερ Σμιτ ήταν απόν στην ψηφοφορία, είχε ψηφιστεί, ζητά να ξαναμπεί στην ημερήσια διάταξη. Έγινε, θα είναι σκόπιμο ίσως, θα ήταν σκόπιμο ωστόσο, να ακούσουμε τον κύριο Μέσσερ Σμιτ πρώτα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Δεν θα πάρω πολύ χρόνο από εσά γιατί ψηφίζουμε. Πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα για το θέμα της διαφάνειας και της δημοκρατίας προχωρούμε προς τις ευρωεκλογέ ε, έξι μήνες. Πολλοί ψηφοφόροι έχουν λογικά αιτήματα να μπορούν να ελέγχουν τον τρόπο με τον οποίο εμείς δρούμε ως πολιτικοί. Ξέρω βεβαίως ότι το Κοινοβούλιο υπερψήφισε, ζήτησε, έχει ψηφίσει πάρα πολλές φορές. Το να ζητάμε ονομαστική ψηφοφορία ίσως είναι πολύ για όλα, αλλά ίσως αρκεί να έχουμε στι τελικές ψηφοφορίε. να υπάρχει ονομαστική ψηφοφορία στις επιτροπέ και στην Ολομέλεια για τις τελικές ψηφοφορίε. Και οφείλω να σα πω ότι με τις, μετά από συζητήσεις που είχα δεν ξέρω γιατί οι σοσιαλιστές αντιτίθενται στην ιδέα αυτή. Πολλοί σοσιαλιστές και συντηρητικοί άλλωστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν να γνωρίζουν ότι οι βουλευτέ που ψηφίζουν τηρούν και σέβονται και τις ε, υποχρεώσεις τους και θέλουν να ξέρουν πώς ψηφίζουν. Ελπίζω αυτό να περάσει και ε, στο πνεύμα της τροπολογίας μου θα ήθελα η ψηφοφορία αυτή να γίνει με ονομαστική ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Μισό λεπτό να δούμε αν πρέπει να δοθεί απάντηση. Κύριε Ντάφ. Ένα τέταρτο των παρόντων πρέπει να υποστηρίξει το αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας. Οι φιλελεύθεροι το υποστηρίζουν και οι πράσινοι το υποστηρίζουν. Και οι συντηρητικοί το υποστηρίζουν. Άρα ψηφίζουμε ονομαστική ψηφοφορία Άρχεται η ψηφοφορία. Όχι, όχι, μισό, δεν είμαστε έτοιμοι. Κύριε Γκουαλτιέρη. Είστε έτοιμοι. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Allora, hanno votato a favore 20, 17 su 24. Ψήφισαν 17, καταψήφισαν 7. εγκρίνεται το κείμενο. Το πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει να το παραπέψουμε στην Ολομέλεια και δεν υπάρχει εισηγητής. Ίσως ο πρόεδρος θα πρέπει να κάνει την... να αναλάβει την έκθεση. Είναι πανευτυχής ο κύριος Μέσσεσμιτ. Λάμπει το χαμόγελό του. Να κάνω εγώ την έκθεση στην Ολομέλεια. Εντάξει. Επόμενο σημείο. Έκθεση για τερμαϊκή. Τροποποίηση του άρθρου 7 του κανονισμού για τις διαδικασίες σχετικά με την άρση και υπεράσπιση της βουλευτικής ασυλίας. Ξεκινάμε. Ψηφίζουμε ομού τις τροπολογίες 16 δικές μας και μία της νομικής που είναι ταυτόσημες υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1 της εισηγήτριας υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Κλείνει το μικρόφωνο. Η τροπολογία 2 αποσύρθηκε. Άρθρο 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 18 ψηφίζουμε. Μετά την 19 που είναι ίδια με την 7 της Γιούρη. Ψηφίζουμε πρώτα την τροπολογία 19 και 7 της νομικής. Καταλάβατε, ψηφίζουμε την 19 της Επιτροπής μας, Βίλεντ Γκαργκάνη και 7 της Γιούρη, υπέρ. 13, 14, 15. 15. 15 favore, contrari. Κατά. Αποχές. Μία αποχή. Εγκρίνονται. Καταπίπτει η 18. Γιατί είναι αντίθετη με αυτά που αναφέρονται εδώ. Τρία της εισηγήτριας και τρία της Γιούρι. Ίδιες. Υπέρ. κατά, αποχές, εγκρίνεται, εγκρίνονται. Τροπολογία 4 της εισηγήτριας και 4 της νομικής. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτές. Τροπολογία 5. 5 είναι και για τη Γιούρη και για την εισηγήτρια. Υπέρ, δύο οι τροπολογίε. Κατά, αποχές δεκτές. Έξι της εισηγήτριας και υπέρ, Κατά. αποχές εγκρίνεται 14 προς 10 τροπολογία 7 αποσύρθηκε 19 ψηφίστηκε τροπολογία 8 της εισηγήτριας και 8 της νομικής υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 της εισηγήτριας Η 28 εγκρίθηκε. ΠΕΡ για την 9 κατά αποχές εγκρίνεται. Η έγκριση του 9 οδηγεί σε κατάπτωση της τροπολογίας 20 Βίλαντ Γκαργκάνη και 9 της Γιούρη. Τροπολογία 10. 10 της ηγήτριας και 10 της νομικής. Υπέρ. Κατά. Ε, αποχές εγκρίνεται. Εγκρίνονται. Τροπολογία 11. Της εισηγήτριας και 11 της νομικής. Υπέρ. 12 της εισηγήτριας υπέρ Κατά. Αποχές. Κανείς. Εγκρίνεται. Άρα καταπίπτει η τροπολογία 12 της νομικής επιτροπής. Τροπολογία 13 της εισηγήτριας που είναι ταυτόσιμο με τις 13 της νομικής υπέρ των δύο τροπολογιών κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 14 της νομικής και 14 της εισηγήτριας. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 15 και τις συγκήτριας και τις νομικής υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 Γκαργάνι Βίλαντ και 16 νομικής ταυτόσημες τροπολογίες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Αιτιολογική σκέψη α με τοποποίηση της συγκήτριας αλλά αποσύρθηκε. Ψηφίζουμε την έκθεση συνολικά. Πρόεδρε. Παρακαλώ να κάνουμε αυτά που λέμε. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά αν γίνεται. Υπάρχει κάποιος που αντιτίθεται. Κι άλλη νίκη του κύριου Μέσσερ Σμιτ. Χριστούγεννα, ο Άι Βασίλη σας έφερε του κόσμου τα δώρα κύριε Μέσσερ Σμιτ. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Με 22 ψήφους υπέρ και μία κατά. Συγχαρητήρια κύριε Γιατερμέκη. Τελειώσαμε με τις ψηφοφορίες. Vabbè, comunicazioni sui coordinatori. Sì, eh, stavo lavorando. tutto. Procederò successivamente Θα σα ε, ενημερώσω κατόπιν για τι ανακοινώσει ε, και συστάσει των συντονιστών. Για να μην ξεχάσω τίποτα, πήραμε κάποιες αποφάσεις, σε ό,τι αφορά του εισηγητές, αλλά θέλω με βοηθήσει η γραμματεία να τα γράψω, ούτω ώστε να μην ξεχάσω τίποτα. Προχωράμε. Εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας, σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο κύριος Ράγκελ μας ενημέρωσε. Έχουμε ένα σχέδιο έκθεση σήμερα του συναδέλφου. Κοιτάξτε, μπορείτε να σταματήσετε να συγχαίρετε τον κύριο Μέσσερ Σμιτ πια. Φτάνει. Ούτε με ακούνε, ούτε με καταλαβαίνουν. riprendiamo con tranquillità il nostro lavoro. Να ξαναρχίσουμε να κάνουμε καμιά δουλειά. Σημείο 14. Applicazione del Trattato di Lisbona. Εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας, λέω. Ο κύριος Άγγελ το, έχει το λόγο. Ε, Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, έχετε την τελική έκδοση του σχεδίου έκθεσης που έχω συντάξει για την εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπως προβλέπει η συμφωνία, στην οποία καταλήξαμε με τους συναδέλφους και τους άλλους βουλευτές, αυτό που θα εξετάσουμε κυρίως είναι οι σχέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο στόχος της έκθεσης αυτής είναι να καλύψει ένα περιορισμένο πεδίο εφαρμογή των σχέσεων της Κομισιόν και του Κοινοβουλίου. Και αυτό αντικατοπτρίζει την διαρθρωτική συμφωνία που είχαμε εδώ στο Κοινοβούλιο. Κάποιοι άλλοι θα εξετάσουν τις σχέσεις με το Συμβούλιο, κάποιοι τις σχέσεις με την Κομισιόν. Ουσιαστικά, αυτό που θα προσπαθήσω να κάνω είναι πάρα πολύ σύντομα να σας ε, παρουσιάσω ε, το αντικείμενο. Δεν ε, υπάρχουν σημαντικές αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη μου παρουσίαση. Σας είχα παρουσιάσει τις αντρές γραμμές την προηγούμενη φορά. Σας παρουσίασα προφορικά τις σκέψεις μου. Δεν μπορώ να πω ότι έχουμε καινοτομήσει έκτοτε ιδιαίτερα, οπότε τι μπορώ να σας πω σήμερα. Πρώτα απ' όλα ότι υπάρχουν δύο μείζονες ε, ανησυχίες, δύο μελήματα. Πρώτον, πώς ενδυναμώσουμε τη δημοκρατική νομιμοποίηση των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων και της Κομισιόν. Και δεύτερον, τα κριτήρια που θέλουμε να εφαρμόσουμε σε ό,τι αφορά την διάκριση εξουσιών. Να υπάρχει κάποια αυστηρότερη διάκριση εξουσιών, διότι στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα ε, το πρόβλημα ίσως να μην έγινε τόσο στη δημοκρατική νομιμοποίηση αυτή καθ' αυτήν, αλλά περισσότερο στις δυσκολίες επίτευξης αυτής της διάκρισης των εξουσιών από νομικής και ουσιαστικής πλευράς προσπαθούμε να πετύχουμε τη διάκριση των εξουσιών. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τους δυτικούς πολιτισμούς, αλλά και σε άλλες ε, περιοχές του κόσμου. Θέλουμε λοιπόν ε, τη διάκριση των εξουσιών ε, να την συμπεριλάβουμε και σε αυτό το εντό αγωγικών ευρωπαϊκό σύνταγμα, αν μπορεί να το πει κανείς. Ενίσχυση λοιπόν δημοκρατικής νομιμοποίησης αφενός και ενίσχυση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών αφετέρου. Αυτή είναι η βασική άξονες του σχεδίου αυτού. Πρέπει επίσης ε, να ε, διευκρινίσουμε και τα της εντολής του καθεθεσμικού οργάνου. Η έκθεση υποδηρείται σε τέσσερα κεφάλαια. Το πρώτο αφορά την νομιμοποίηση και την πολιτική ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και εκεί θίγεται και το θέμα του ορισμού του Προέδρου και των Επιτρόπων. ή τη δυνατότητα συζητάμε να ε, αποπεμφθούν από, την, ε, από το σώμα των επιτρόπων με πρόταση ή με κάποιο άλλο τρόπο κάποιοι επίτροποι. Επίσης, νομοθετική πρωτοβουλία, δραστηριότητες για την πρόθεση νομοθετημάτων από το Σκηνοβούλιο και από την Κομισιόν. Ή κάτι άλλο που εξετάζουμε είναι Ποιο είναι ο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην πρόταση ε, νομοθεσία αλλά και στην άσκηση δημοκρατικού ελέγχου ε, πάνω στην ε, πρωτοβουλία που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να νομοθετεί. Και άλλο πώ ασκούμε και πλήρω τον κοινοβουλευτικό μα έλεγχο επί των εργασιών τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, όπω όλοι γνωρίζετε, Υπάρχει το ζήτημα των κατεξουσιοδότηση πράξεων, ε, διότι με τις κατεξουσιοδότηση πράξεων αλλάζει το σκηνικό. Η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων ε, πραγματεύεται το θέμα αυτό. Ε, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, περιεκτικός, αλλά δυστυχώς θα είμαι πιο περιεκτικός από όσο θα έπρεπε για να μπορέσω να περάσω σωστά τα μηνύματα. Θα δούμε και το θέμα των διεθνών σχέσεων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εφηγραμμίζει τις πρωτοβουλίες και τις αρμοδιότητές του με το σωστό τρόπο. Θα δούμε και τα συνταγματικά ζητήματα που αφορούν τις διοργανικές συμφωνίες. Αυτές οι συμφωνίες βασίζονται στη συνθήκη της Λισαβόνας. Αυτή είναι η συνταγματική βάση, αν θέλετε, το χειρώνεται στις συνθήκες. Αλλά αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε στην εκθεσή μας είναι κάνουμε ένα είδος πρόβλεψης, πρόγνωσης, να εκτιμήσουμε κάπως την κατάσταση, βλέποντας πώς έχουν εξελιχθεί οι σχέσεις μεταξύ Κομισιόν και Ευρωκοινοβουλίου μέχρι τώρα και να δούμε στο μέλλον ε, τι μορφή θα μπορούσαν να έχουν αυτές οι σχέσεις και τι θα μπορούσε να είναι το περιεχόμενο μελλοντικών διοργανικών συμφωνιών. Είπαμε ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να συμμετέχει στις διαδικασίες και το Συμβούλιο, αλλά θα πρέπει η εντολή, οι αρμοδιότητες του κάθε οργάνου να γίνονται σεβαστές η δυνατότητα διμερών ε, συμφωνιών μεταξύ Κοινοβουλίου και Επιτροπής είναι μια άλλη δυνατότητα. Εκεί δεν θα πρέπει να παρεμβαίνει το Συμβούλιο, γιατί έχουμε αυτή την ε, αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Προσπαθούμε λοιπόν να οργανώσουμε με κάποιος, κάπως συστηματικό τρόπο την έκθεση αυτή γύρω από τέσσερις πυλώνες. Επίσης ε, επειδή έχω κάνει ήδη προφορική παρουσίαση της έκθεσης ε, και επειδή έχετε μπροστά σας τώρα την έκθεση, δεν ξέρω αν είχατε χρόνο να την ε, διαβάσετε. Πότε τη λάβατε αυτή την έγγραφη εκδοχή σήμερα το πρωί, δεν ξέρω. Είχατε χρόνο να την κοιτάξετε, αλλά ε, αν όχι, ίσως θα μπορούσα να σας αναφέρω τα πιο σημαντικά στοιχεία της έκθεσης. Πρώτα απ' όλα, νομιμοποίηση, πολιτική ευθύνη θα ήθελα να, εφιστήσω, να επιστήσω συγγνώμη την προσοχή σας στο ότι το ουσιώδες εδώ είναι με ποιο τρόπο το εκλογικό σώμα θα βλέπει τις επιλογές του να αντικατοπτρίζονται στο έργο της Κομισιόν. Και μιλώ ιδίως εδώ για την εκλογή, τον ορισμό του Προέδρου της Κομισιόν και των Επιτρόπων. Γνωρίζουμε ότι έχουν επέλθει αλλαγές ε, ώστε τα πολιτικά κόμματα να μπορούν να έχουν λόγο ε, στην υποψηφιότητα και στο ποιος τελικά θα οριστεί ω πρόεδρος τη Κομισιόν. Πώ όμως οι ψηφοφόροι μπορούν να επηρεάσουν ευρύτερα το πολιτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για κάτι τέτοιο θα πρέπει και το Κοινοβούλιο ε, φυσικά να έχει έτοιμο το πρόγραμμα του πριν τις εκλογές, αλλά και το Συμβούλιο ε, θα πρέπει να δούμε πώς θα ανταποκρίνεται στις επιλογές του Κοινοβουλίου ή των πολιτών. Και όταν οριστεί ο πρόεδρος της Κομισιόν, τι θα γίνει με τους ε, επιτρόπους, πώς θα ορίζονται αυτοί. Έχουμε ακούσει τη λεγόμενη μαξιμαλιστική προσέγγιση, υπάρχει και σε ένα επεξηγηματικό σημείωμα, αλλά εμείς θέλουμε να υπάρχει ισορροπία μεταξύ κοινοβουλευτικού ελέγχου να μην έχουμε υπερβολική βέβαια ε, κοινοβουλευτική παρέμβαση και εκεί εστιάζω και την προσοχή μου. Από τότε που έγινα βουλευτής ε, θεωρούσα ότι ε, για να είμαστε αποτελεσματικοί πρέπει να είμαστε ενεργοί, δραστήριοι, όχι όμως υπερβολικά. Πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί οι βουλευτές του Κοινοβουλίου. Ίσως κάποιες φορές ορισμένοι δεν αντιλαμβάνονται είτε τη συνταγματική ιστορία των κρατών μελών, ε, κάποιες φορές ε, προωθούν κάποια πράγματα ή αντιδρούν σαν να ε, έχουμε μια κοινοβουλευτική ιστορία διαφορετική. Δεν θα πρέπει να προσπαθεί το κοινοβούλιο να αντικαταστήσει την κυβέρνηση ούτε σε εθνικό επίπεδο, άρα και εδώ στο ευρωπαϊκό επίπεδο δεν θα πρέπει να προσπαθεί το Κοινοβούλιο να αντικαταστήσει την Κομισιόν, θα πρέπει να ασκεί έλεγχο, θα πρέπει να έχει περιθώρια αυτονομίας κινήσεων, θα πρέπει να υπάρχει μια σωστή διάκριση εξουσιών Και το άρθρο 16 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ξεκάθαρα προβλέπεται θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα δικαιώματα των πολιτών, αλλά να υπάρχει διάκριση των εξουσιών. Σίγουρα βέβαια η άσκηση ελέγχου δεν θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την παρακόλληση της ανάληψης δράσης από την Κομισιόν. Σίγουρα ο πρόεδρο τη Κομισιόν θα πρέπει να έχει κάποια αυτονομία στην επιλογή των επιτρόπων για να μπορεί να δουλεύσει σωστά η Κομισιόν. Είχαμε προτείνει μια λίστα τριών επιτρόπων, από του οποίου θα επιλέγει έναν ο πρόεδρο τη Κομισιόν. Και τα κράτη-μέλη μπορούν, επαναλαμβάνω, να προτείνουν ένα κατάλογο με τρία, τρει υποψηφιότητε. Και βέβαια λαμβάνοντα υπόψη και την ισορροπία μεταξύ των δύο φύλων. Και αυτό είναι κεντρικό σημείο. Τώρα, για να εξασφαλίσουμε την ανεξαρτησία της εκτελεστικής εξουσίας, να έχει τη δυνατότητα να ενεργεί, να δρά. Και σε επεξηγηματικό σημείο θα το δείτε αυτό πάλι. Δεν μπορούμε να το βάλουμε στο σώμα της έκθεσης, είναι σε ένα επεξηγηματικό σημείο. Θεωρούμε ότι ο ρόλος ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποδυναμώνεται. Πώς μπορούμε λοιπόν να τον ενισχύσουμε, πώς μπορούμε να ενδυναμώσουμε την Κομισιόν ναι, να εναμιγήσω ο ρόλο. της. Πρώτα απ' όλα, θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε τη δημοκρατική της νομιμοποίηση. Και αυτό πώς μπορούμε να το πετύχουμε, με καλύτερο κοινοβουλευτικό έλεγχο, πρώτο σημείο. Δεύτερο σημείο, μπορούμε να ενισχύσουμε την εκτελεστική αυτονομία, άρα και την αποτελεσματικότητα της Κομισιόν. Αυτό μπορεί να το πετύχουμε δίνοντας περισσότερες εξουσίες, ε, ε, περιθώρια, διακριτική ευχέρεια στην Κομισιόν. Αυτός είναι ο ένας τρόπος. Μια άλλη σημαντική πτυχή βέβαια είναι να γίνει πιο αποτελεσματικό το έργο της Κομισιόν. Ξέρουμε ότι είναι φιλόδοξη συνθήκη της Λισαβόνας. Εκεί προβλέπεται ότι θα έπρεπε να μειωθεί ο αριθμό ε, των επιτρόπων ώστε να καλύπτουν τα δύο τρίτα των κρατών μέλων. Μείωση δηλαδή το ρυθμό των επιτρόπων. Είδαμε όμως ότι αυτό ήταν σφάλμα τελικά. «11 Δεκεμβρίου του 2008» αναφερόταν στην έκθεση μια προθεσμία. Λάθος είναι αυτό. Τέλος πάντων, μετά το δημοψήφισμα στην Ιρλανδία αποφασίστηκε ότι κάθε κράτος μέλος θα συνεχίσει να έχει έναν επίτροπο για την επίλυση του προβλήματος σας πρότεινα μια καινοτόμο, ίσως και επίμαχη λύση, αλλά πιστεύω ότι είναι η μέση οδός, είναι μια χρυσή τομή, ένα συμβιβασμός για την συμφιλίωση των δύο αντικρουόμενων ε, στόχων. Δηλαδή να έχουμε τα δύο τρίτα της Κομισιόν που έχουν χαρτοφυλάκιο, τα δύο τρίτα, τα δύο τρίτα δηλαδή των επιτρόπων που θα έχουν χαρτοφυλάκιο και το ένα τρίτο που δεν θα έχει χαρτοφυλάκιο. Δηλαδή θα πρέπει κανείς να επιλέγει τους επιτρόπους που θα έχουν χαρτοφυλάκιο με βάση ε, τις, ε, τους όρους της Νίκης της Λισαβόνας. Ε, σύστημα εκπεριτροπής, εναλλάσσονται οι χώρες με βάση ε, τα γεωπολιτικά κριτήρια και θα υπάρχουν και άνευ χαρτοφυλακίου επίτροποι με τον τρόπο αυτό προσπαθούμε να ε, αποκαταστήσουμε την ισορροπία μεταξύ μικρότερων, μεγαλύτερων χωρών και ε, να έχουμε μια καλή γεωγραφική κάλυψη, σύμφωνα με τους όρους της συνδίκησης της Λισαβόνας. Όλα αυτά βέβαια θα αποτελέσουν αντικείμενο πολυπλοκότητα των διαπραγματεύσεων. Για να έχουμε πενταετίες όπου θα μπορεί η Κομισιόν να έχει ε, τη δυνατότητα με τα χαρτοφυλάκια να επιτελέσει σωστά το έργο της. Λέμε λοιπόν πρόταση 2 τρίτο των επιτρόπων μετά χαρτοφυλακίου και 1 τρίτο άνευ χαρτοφυλακίου. Και αυτοί οι άνευ χαρτοφυλακίου επιτρόποι τι θα κάνουν τέλος πάντων. Πρώτον θα μπορούν να, να εκπροσωπούν την Κομισιόν. Ακόμη και 200 ημέρες εκτός Βρυξελών ε, παραπονούνται ορισμένοι επίτροποι ότι πρέπει να ε, δαπανούν. Θα μπορούσαν ε, λοιπόν να έχουν μεγαλύτερη ελευθερία αυτοί που έχουν το χαρτοφυλάκι και αυτοί που δεν το έχουν θα μπορούσαν να εκπροσωπούν την Κομισιόν εκτός Ένωση ή και εντός Ένωσης, να μετακινούνται δηλαδή πιο πολύ από τους άλλους. Επίσης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλα τα συμφέροντα να υπάρχει περισσότερη αμεροληψία. Από τότε που σπουδάζαμε, το δικτικό δίκαιο τα μαθαίναμε αυτά. Δεν θα πρέπει να παραγνωρίζουμε τα εθνικά συμφέροντα. Καλό είναι κάπως να τα ε, βάλουμε στο ίδιο καλάθι με τον τρόπο ώστε να προωθούμε συλλογικά συμφέροντα περισσότερο σίγουρα δεν θα κάθονται ε, να άπραγοι ε, όλη τη μέρα αυτή η Επίτροπη Ανευχαρτοφυλακίου. Θα πρέπει και αυτοί να αναλάβουν κάποιες αρμοδιότητες. Αν έχουμε 7-8 επιτρόπους χωρίς χαρτοφυλάκιο, δεν θα μπορούμε να προχωρήσουμε στη μελέτη των ε, διαφορών φακέλων. Δεύτερον, θα με ρωτήσετε, η λύση είναι ιδεώδης, ίσως όχι, αλλά είναι ισορροπημένη και σέβεται τις αρχές της Λισαβόνας και την αντιπροσωπευτικότητα. Κατά την άποψή μου θα ήταν μια ενδιαφέρουσα λύση. Να πω ακόμα κάτι. Μας ανησυχεί ιδιαίτερα το θέμα της δημοκρατικής νομιμοποίησης της Επιτροπής. Προσοχή. Δύο είναι τα βασικά συμφέροντα. Να υπάρξει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, αυτονομία και ελευθερία για την Επιτροπή. Τούτο θα γίνει μέσω, γίνεται μέσω της επιλογής του Προέδρου της Επιτροπής και μία μεγαλύτερη ε, και μιας μεγαλύτερης ε, αποτελεσματικής λειτουργίας επιτρόπων με και χωρίς προϋπολογισμό. Πώς θα γίνει αυτό ευκολότερα μέσω των ευρωεκλογών είναι σημαντικό να ασκηθεί πίεση στο Συμβούλιο ούτω ώστε να αναλάβει το Συμβούλιο να δίνει απαντήσεις στις διαβουλεύσεις που έχουν γίνει μετά την συνθήκη της Λισαβόνας και άρα είναι θεμελιώδες να εξασφαλιστεί κάτι τέτοιο. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό σε μία μελλοντική συνέλευση να μειωθεί το ποσοστό της ε, ειδική πλειοψηφίας για την Επιτροπή. Εμείς έχουμε ειδική πλειοψηφία, όχι απλή ή απόλυτη πλειοψηφία για την ε, πρόταση μομφής κατά της Επιτροπής. Ε, αυτό επιβαρύνει τη θέση του Κοινοβουλίου. Κάτι, άλλη, κάτι άλλο σημαντικό που δεν το θυμούνται, δεν το ξέρουν ίσω οι συνάδελφοι, είναι το εξής. Πρέπει να αναθεωρήσουμε όπως και δίποτε τις δυνατότητες ατομικής ε, πρότασης μορφής. Δηλαδή την υποχρέωση ε, ανάκλησης ενός ατομικού ε, ενός ατομικού επιτρόπου. Ε, αυτό δεν είναι κοινοβουλευτικό. Είναι ε, σύστημα κυβερνώσας βουλής που δεν υπάρχει σε μας. Δηλαδή ίσχυε στη Γαλλία κατά τη διάρκεια της, ε, μετά τη Γαλλική Επανάσταση μεταξύ του 93-95 μετά τη Γαλλική Επανάσταση στην Δημοκρατία. Ε, ελπίζω ότι θα φτάσουμε εκεί, λέει ο συνάδελφο, δίπλα και όντω και εγώ το ελπίζω. Είναι λοιπόν σημαντικό να τονίσουμε το εξή. Οι βουλευτές θέλουμε περισσότερες εξουσίε και μερικέ φορές ζητάμε πράγματα που δεν σέβονται το δημοκρατικό σύστημα. Φερρυπίν. Ε, σε ό,τι αφορά τι διεθνεί συμβάσει, Οι διεθνεί συμβάσει πουθενά δεν είναι αντικείμενο Διαπραγμάτευση από τις βουλές, αλλά από, από την εκτελεστική εξουσία. Στο τέλος, όταν υπάρχει το τελικό κείμενο, ψηφίζεται αυτό το κείμενο από τη Βουλή. Αυτό έλεγε ο Μοντεσκέ. Η διαπραγμάτευση των διεθνών συμβάσεων είναι θέμα της κυβέρνησης, όχι της Βουλής. Δεν μπορεί να πάμε όλοι να κάνουμε διαπραγμάτευση σε διεθνές επίπεδο. Πρέπει να ακολουθήσουμε λοιπόν τα αυστηρά κριτήρια του, της διάκρισης των εξουσιών. Το οποίο είναι στο, πρέπει να μπει στο κέντρο της πολιτικής ζωής της Ευρώπης. Μίλησε τώρα για την συνέλευση, την ανάγκη μείωσης του αριθμού της πλειοψηφίας, την μείωση της ειδική πλειοψηφίας που είναι αναγκαία για να υπάρξει μία πρόταση για να περάσει μια πρόταση μορφής. Ελπίζω αυτό να, μην, να συζητηθεί σε μια επόμενη συνάντηση. Κάτι άλλο σημαντικό είναι να αποφασίσουμε θα προχωρήσουμε προς ένα κοινοβουλευτικό ή ένα προεδρικό μοντέλο. Όπως σας είπα, δεν πρέπει να αποκλείσουμε μια τέτοια, ε, ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Η μία θεσμική δυνατότητα της Ένωση είναι η άμεση εκλογή του Πρόεδρου. Υπάρχουν πλονεκτήματα με, με το μοντέλο αυτό. Ξέρω ότι πολλοί δεν το θέλουν. Να σας πω τα πλονεκτήματα. Το πρώτο είναι ότι μπορούμε να εξισορροπήσουμε τις εξουσίες. Εμείς έχουμε, όπως περιγράφει η έκθεση, την οπτική που υποστηρίζουμε εδώ. Δηλαδή, αύξηση της δημοκρατικής νομιμοποίησης του Κοινοβουλίου και του ελέγχου της Επιτροπής. Στο μέλλον θα έχουμε δηλαδή έναν διεισμό Επιτροπή Κοινοβούλιο που προστατεύουν τα συμφέροντα της Ένωσης, κράτη Συμβούλιο που προστατεύουν τα συμφέροντα των κρατών. Θα υπάρχει μια, μια μάχη μεταξύ δύο νομιμοποιήσεων, της Ευρωπαϊκής αφενός και των κρατών μελών αφετέρου, στην πράξη θα αποτελούν τους δύο συγκρούμενους άξονες. Αν υπήρχε προεδρικό σύστημα, όπου ο πρόεδρος της Επιτροπής εκλέγεται από τους πολίτες, αυτό είναι ένα μοντέλο, η τάση θα ήταν να γίνει το Συμβούλιο μια δεύτερη βουλή, μια άνοβουλή που θα επέτρεπε να αποφύγουμε τον κίνδυνο συνταγματικής σχιζοφρένειας, όπου θα υπάρχει ένα θεσμικό όργανο που λειτουργεί σαφώς στην διακυβερνητική δια, δια, ε, λογική και εκπροσωπεί τα κράτη-μέλη και δύο θεσμικά όργανα που θα επιδιώκουν τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Με το προεδρικό σύστημα χάνεται η σχιζοφρένεια αυτή. Ξέρω ότι το σύστημα αυτό έχει και ένα άλλο πλεονέκτημα. Δείτε περιπτώσεις της Ινδίας, του Καναδά, όπου χρησιμοποιείται τέτοιο σύστημα. Μα τι... Στην Ινδία υπάρχει προεδρικό σύστημα, για παράδειγμα. αυτό θα έχει επιπτώσεις. Δεν θα υπάρχει κοινοβουλευτική επίπτωση στην Επιτροπή και ίσως θα πρέπει να φύγει, δηλαδή θα έχει λόγο ύπαρξη, η πρόταση μομφής. Θα μπορούσαμε ίσως να διακρίνουμε, να διατηρήσουμε μια ατομική πρόταση μομφής. Τέλος πάντων, αυτά δεν τα λέει η έκθεση. Η έκθεση λέει ότι στην συνέλευση πρέπει να σκεφτούμε να δώσουμε μεγαλύτερη δημοκρατική νομοποίηση στην Επιτροπή και να μην αποκλείσουμε, δεν λέει αποθαρρύνουμε, το ενδεχόμενο να προχωρήσουμε προς ένα προεδρικό σύστημα και όχι αυτή τη ε, κοινοβουλευτική ε, προσέγγιση που υποστηρίζει η έκθεση. Εγώ δεν έχω προηλημένε θέσει μεταξύ των διαφόρων μοντέλων. Ωστόσο, πιστεύω ότι στη φάση αυτή θα έπρεπε να σταθούμε περισσότερο στην, στην ε, κοινοβουλευτική διάσταση. Προτείνω γιατί. Πρώτον, αυξάνει την δημοκρατική νομιμοποίηση και δεύτερον αυξάνει, δεύτερον τον έλεγχο του Κοινοβουλίου και τρίτον ενισχύει την αυτονομία της εκτελεστικής εξουσίας ενισχύοντας την διάκριση των εξουσιών. Είναι θεμελιώδη αυτά τα τρία σημεία. Ενισχύουμε την νομιμοποίηση της Επιτροπής μέσω των εκλογών και της ευκολότερης πρότασης μορφής. Δεύτερον, ε, διευκολύνουμε την, το δημοκρατικό έλεγχο του Κοινοβουλίου. Την υποχρέωση, για παράδειγμα, του υποψήφιου Προέδρου του Συμβουλίου να, να έρχεται, όπως έκανε στη θυμή αυτή, να παρουσιάσει τους βασικούς προσανατολισμούς και το πρόγραμμά του πριν λάβει την ψήφο του Κοινοβουλίου. Και τρίτον, το ετήσιο πολιετές πρόγραμμα, το ετήσιο πρόγραμμα ε, της, ε, νομοθετικό πρόγραμμα της Επιτροπής θα πρέπει να την χάνει της επικύρωσης του Κοινοβουλίου. Αυτό ενισχύει την ε, επιρροή του Κοινοβουλίου που πρέπει να, να συμπληρωθεί από την άλλη πλευρά του νομίσματος, όχι την άλλη πλευρά του, της Ελλήνης, γιατί ποτέ δεν τη βλέπουμε. Το, η άλλη πλευρά του νομίσματος είναι η αυτονομία της εκτελεστικής εξουσίας, ενισχύοντας τις δυνατότητες επιλογής ε, των ε, επιμέρους επιτρόπων με μεγαλύτερη διακριτική ευχαίρεια από πλευράς πρόεδρου της Επιτροπής. Αυτά. αυτή είναι η δρόμη μέσω των οποίων υλοποιείται και συγκεκριμενοποιείται η νομοποίηση της Επιτροπής. Επίσης, να σας, επιστήσω, να σας επιστήσω την προσοχή στην νομοθετική δραστηριότητα. Α, κάτι ξέχασα. Σημαντικό. Το εξής. Όταν ζητήσαμε από τον πρόεδρο της Επιτροπής να παρουσιάσει το πρόγραμμά του πριν ψηφιστεί, για να ενισχυθεί η παρέμβαση του Κοινοβουλίου στην επεξεργασία του ετήσιου νομοθετικού και του πολιετούς νομοθετικού προγράμματος της Επιτροπής. Ακολουθούμε αντικειμενικά κριτήρια. Το ξαναλέω. Ακολουθούμε αντικειμενικά κριτήρια. Για να ξέρουμε ποια σημεία είναι σημαντικά για μας και πού μπορούμε να παρέμβουμε. Σε πολλές περιπτώσεις νομοθετικά κείμενα πέρασαν με 500 και 600 ψήφους ε, στο Κοινοβούλιο χωρίς να γνωρίζουμε ωστόσο, χωρίς να έχει υποβληθεί πρόταση από την Επιτροπή στο ετήσιο προγραμματισμό. Προτείνω λοιπόν όταν η Επιτροπή αποφασίζει για τα ετήσια προγράμματα θα πρέπει να λάβει υπόψη την μεγάλη συνένεση που ακολουθεί, που έχει το Κοινοβούλιο για θέματα περί Φερρυπίν της ψηφιακής ενιαίας αγοράς ή της εμβάθυνσης της ε, ενιαίας αγοράς ή της αγοράς ενέργειας ή τα άλλα των άλλων βασικών θεμάτων για την ε, τραπεζική ή την οικονομική ένωση, θέματα δηλαδή που είχαν μαζική συνένεση στο Κοινοβούλιο που υποστηρίχθηκαν από πολλές και όλες σχεδόν τις πολιτικές ομάδες και που η Κομισιόν αγνοεί παντελώς τώρα. Έχουμε αντικειμενικά κριτήρια που μπορούν να εμπνεύσουν τους βουλευτές της Νέας Φοιτείας για να προχωρήσουν δίνοντας ένα πολιτικό περιεχόμενο στο πρόγραμμα του Πρόεδρου της Επιτροπής. Διότι η Επιτροπή πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ψηφοφορίες στο Κοινοβούλιο και τούτο να είναι γνωστό τη στιγμή της έγκρισης του Πρόεδρου. Θα μου πει κάποιος, αυτό δεν είναι εκβιασμός. Όχι. Ξέρουμε ότι πολλά κοινοβούλια, η Βρετανία για παράδειγμα, δείχνουν ότι σε πολλές περιπτώσεις η Βουλή υποχρέωσε κοινοβούλιο να δεχθεί, η υποχρέωση την κυβέρνηση να δεχθεί με την απειλή του impeachment ενδεχόμενα την ε, αύξηση των εξουσιών του. Είναι εργαλεία ενίσχυση της δημοκρατίας αυτά. Προφανώ η απόφαση αυτή δεν θα είναι απόφαση του τωρινού κοινοβουλίου, αλλά ίσως του επόμενου, αυτού που θα εκλογεί το Μάιο του 2014. Έχουμε ωστόσο κι εμείς ένα track record, έχουμε το μητρό της δράση μας στο παρελθόν. Σε ό,τι αφορά την νομοθετική δραστηριότητα θα σας πω το εξής. Πολλά πρέπει να δούμε. Το πρώτο στο οποίο πρέπει να σταθούμε είναι να δουλέψουμε για μια συνέλευση, αλλά και πέραν της συνέλευσης να δουλέψουμε για διοργανικές συμφωνίες, ούτως ώστε να αποκτήσει το Κοινοβούλιο το δικαίωμα της νομοθετικής πρωτοβουλίας. Καταλαβαίνω ότι στο πλαίσιο των checks and balances, των ελέγχων και ισορροπιών της ευρωπαϊκής πολιτικής ζωής, η νομοθετική πρωτοβουλία, η αποκλειστική νομοθετική πρωτοβουλία της Επιτροπής είναι το τελευταίο προπίδιο της εξουσίας της. Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή η Επιτροπή είναι διχασμένη ανάμεσα στην μάχη εξουσίας μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Εάν εμείς τις αφαιρέσουμε την νομοθετική πρωτοβουλία, αποδυναμώνεται η Επιτροπή. Αλλά θα, εγώ ζητώ να αυξηθεί η νομοθετική, ε, η δημοκρατική νομοποίηση της Επιτροπής και πιστεύω για να καλύψουμε ακριβώς το έλλειμμα ε, δημοκρατίες Και άλλωστε μην ξεχνάτε ότι ένα κοινοβούλιο χωρί νομοθετική πρωτοβουλία είναι ανήκουστο. Είτε με άμεση πρωτοβουλία μπορεί να γίνει αυτό, είτε μέσω πρωτοβουλία πρωτοβουλίας που έχουμε με άτυπο τρόπο σήμερα. Να ζητά δηλαδή το Κοινοβούλιο από την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει την νομοθετική της πρωτοβουλία ε, σε μια τέτοια περίπτωση η Επιτροπή θα πρέπει είτε να το κάνει είτε να δικαιολογήσει γιατί δεν το κάνει. Αυτό επινισχύει την ε, νομοθετική πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου. Προφανώς εδώ τα θέματα είναι πολλά και ακούω και βλέπω και τον κύριο Μπρόκ δίπλα που κουνιέται στην καρέκλα του γιατί περιμένει να μιλήσει το ξέρουμε όλοι. Λοιπόν, να συνοψίσω. Η, νομοθετική, η συνήθις νομοθετική πρωτοβουλία περιλαμβάνει πολλά πράγματα. Γεωργία, αλληλεία, ενιαία αγορά. Αυτό είναι σημαντικό συνάδελφοι, το ξέρουμε. Το ξέρουμε από το εθνικό πλαίσιο. Σε ορισμένε περιπτώσεις πρέπει να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα των κρατών, των κυβερνήσεών μας και δεν έχουμε επαρκή ενημέρωση. Τι συμβαίνει τώρα στη νομοθετική πρωτοβουλία. Πολλές φορές το Συμβούλιο έχει πρόσβαση σε πληροφορίες πολύ νωρίτερα από εμά. Αυτό δημιουργεί μία de facto ασυμμετρική σχέση μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου που είναι και τα δύο νομοθετικά όργανα. Πρέπει λοιπόν αυτή η προνομοθετική φάση να αποκτήσει μεγαλύτερη ισορροπία. Δηλαδή, οι πληροφορίες που δίνονται στο Συμβούλιο να δίνονται παράλληλα και στο Κοινοβούλιο. Είναι αναγκαίο να... Δείχνει ότι δεν είναι ικανοποιημένο, διακόπτει ο πρόεδρο. Θέλει να, να σας πάρει το λόγο ή πρέπει να φύγει. Αν γίνεται κύριε συνάδελφε να συντομεύετε. Έλεγα λοιπόν ότι υπάρχει και αυτή η διάσταση. Η ασυμμετρία ενημέρωσης των δύο νομοθετικών οργάνων. Υπάρχουν και άλλες ε, σημαντικές ε, παράμετροι. της πράξης, για παράδειγμα. Και εκτελεστικές πράξεις. Για μας αυτό είναι σημαντικό θέμα. Ο Σάγερ έχει κάνει μια πληρέστατη δουλειά για το θέμα αυτό από την νομική επιτροπή. Δεν θέλω να σταθώ περισσότερο σε αυτό. Έχει και νομοτεχνική και συνταγματική διάσταση το θέμα. Άρα πρέπει να, να απασχολήσει και εμάς. Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, διότι οι συνταγματικές εξουσίες που δίνει η συνθήκη αλλοιώνονται από την κακή χρήση των κατεξουδότηση και των εκτελεστικών πράξεων. Είναι σαφές ότι το θέμα της επιτροπολογίας, όπως είναι γνωστή αυτή η διαδικασία, μπορούν να αντιμετωπιστούν το μελλοντικό framework agreement. Πρέπει να φύγει ο κύριος Μπροκ. Να διακόψουμε λίγο αυτά που μας λέτε. Εντάξει. Ο κύριος Μπροκ. Ναι, θα ήθελα να στήσω συγγνώμη από τον συνάδελφο Ρανζέλ, αλλά περιμένω και με περιμένει μάλλον ο εκπρόσωπος της ε, Επιτροπής Ενωμένων πολιτείων στο γραφείο μου και τον έχω στήσει και όλα 10 λεπτά. Λοιπόν, σας σα ευχαριστώ πολύ, κύριε Σίγητά. Θα ήθελα και εγώ να πω δύο λόγια. Εγώ θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική την έκθεση αυτή, διότι μας δίνει τη δυνατότητα να αποφασίσουμε πλέον και να αποφασίζουμε μάλλον για τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό είναι στρατηγική σημασία σε εξέλιξη. Και πιστεύω πως ε, είναι κάτι που πρέπει να γίνει οπωσδήποτε. Πιστεύω πως ο συνάδελφος κύριος ε, Ράνιελ έχει κάνει μια σειρά πάρα πολύ καλών και σημαντικών προτάσεων. Εντάξει, μπορούμε να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες, τα επιμέρους σημεία, ενδεχομένως υπάρχουν μερικές διαφωνίες, όμως οι γενικές γραμμές ε, είναι πάρα πολύ καλή και θέλω να επικεντρωθώ σε ορισμένες ε, συνταγματικής εφήσεως πτυχές. Καταρχάς πιστεύω ότι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ε, ε είναι σε τον οποίο μπορούν, την υποψηφιότητα του οποίου να μπορούν να αρνηθούν εάν δεν θεωρούν πως είναι κατάλληλος. Αυτό βέβαια θα σημαίνει τα κράτη-μέλη στο μέλλον να μην είναι υποχρεωμένα μόνο να ορίσουν έτσι κάποιον που πολλές φορές θεωρούν πως είναι πολιτικός δεύτερης τάξης, αλλά πραγματικά να βρουν κάποιον ικανό για την θέση αυτή. Επίσης, αριθμός των επιτρόπων. Εγώ πιστεύω πως 14 είναι αρκετοί. Οι υπόλοιποι θα μπορούσαν να είναι επίτροποι χωρίς χαρτοφυλάκιο, με δικαίωμα όμως ψήφου. Επίσης, πιστεύω πως η αρχή του ανασχηματισμού είναι πάρα πολύ σημαντική στις, ε, στα χαρτοφυλάκια των επιτρόπων. Θα, πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ένας ε, επίτροπος να αντικαθίσταται από κάποιον άλλον. Δεν πρέπει να υπάρχει δηλαδή η απόλυτη ελευθερία και ένας επίτροπος να νομίζει ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Όχι, πρέπει να υπάρχει αυτή η πίεση ε, της ε, αναπάσα στιγμής αντικατάστασης αν δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Και πιστεύω πως αυτό το εργαλείο πίεσης είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο, διότι με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η ισορροπία. Η ισορροπία μεταξύ μεγάλων και μικρών χωρών και κατά συνέπεια η δημοκρατία. Επίσης, όσον αφορά την πρόταση μομφής, Εγώ, όπως και στα εθνικ στις εθνικές κυβερνήσεις ε, γίνεται αυτή η πρόταση μομφής και κάποιος υπουργό είναι υπόλογος για αυτά που κάνει. Εδώ δεν συμβαίνει μέχρι τώρα κάτι τέτοιο. Και πρέπει να υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Επίσης, ένας ε, επίτροπος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ορίζει ο ίδιος το γενικό του διευθυντή, όπω ακριβώ και σε ένα υπουργείο, σε μια εθνική κυβέρνηση, να ορίζει τον ε, γενικό διευθυντή της, ε, του τμήματό του και να μπορεί και να τον απολύει αν δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Υπάρχει πολιτική ευθύνη. Και αυτή η πολιτική ευθύνη δεν είναι κάτι που απολαμβάνεται πλήρως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τώρα. Οι γενικές διευθύνσεις αντίθετα κατευθύνουν τους επιτρόπους και όχι οι επίτροποι τις γενικές διευθύνσεις τους. Αυτό ε, τώρα όσον αφορά το Συμβούλιο. Και εδώ ισχύουν πάνω κάτω τα ίδια. Εδώ έχουμε στους ε, τριμερείς διαλόγους εκλεγμένους αντιπρόσωπους. Εμάς, όμως, δεν έχουν όλες οι πλευρές ε, την ίδια διαπραγματευτική δυνατότητα, τις ίδιες διαπραγματευτικές αρμοδιότητες και πρέπει να επέλθει ισορροπία στους ετριμερείς διαλόγους. Να υπάρχουν υπουργοί εκλεγμένοι και όχι κάποιοι δημόσιοι υπάλληλοι. Και πραγματικά η κατάσταση αυτή έχει φτάσει στο μη περαιτέρω. Έχουμε ευθύνες που και αρμοδιότητες που προκύπτουν από τις συμβάσεις. Αναφέρεται ένα συμβούλιο, όχι πολλά συμβούλια υπουργών. Θα πρέπει φυσικά να αλλάξει και ο εσωτερικός κανονισμός του Συμβουλίου, έτσι ώστε το Συμβούλιο να γίνει δεύτερη βουλή, μια άνω βουλή. Και αυτό προς το παρόν είναι ένα από τα κυριότερα προβλήματα που έχουμε. Δεν υπάρχει γενική ευθύνη στις πράξεις των Υπουργών και υπάρχει μεγάλη διαφορά σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Εάν όμως υπάρχει επίσημη συναπόφαση Συμβουλίου και Κοινοβουλίου ως δύο βουλές, τότε δεν θα μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να υπεκφεύγουν και να ε, αρνούνται τις ευθύνες τους. Θα έχουν πλέον τις ίδιες ευθύνες με το Κοινοβούλιο και δεν χρειάζεται να αλλάξουν οι συνθήκες για να γίνει κάτι τέτοιο. Τώρα, επίσης, όσον αφορά την, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να πω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι εδώ για να κάνει μικροδιαχείριση και αυτές τις ε, ε μικροδουλειές και εδώ συμφωνώ με τον ε, συνάδελφο κύριο Ραντζέλ. Δεν πρέπει το Κοινοβούλιο να διεξάγει διαπραγματεύσεις Πρέπει να υπάρχει ένα σαφής διαχωρισμός. Να υπάρχει επιρροή βέβαια του Κοινοβουλίου, αλλά να μην αναλαμβάνει το Κοινοβούλιο όλες ε, αυτές τις ε, λεπτομέρειες. Ε, και αυτό είναι συνταγματικά λάθος πιστεύω. Είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όχι ενός Κοινοβουλίου. Και ένας επίτροπος δέχεται πάρα πολλές επιέσεις για τις αποφάσεις που παίρνει. Γι' αυτό πιστεύω πως πρέπει να βρεθεί μία λύση. Και... πρέπει να υπάρξει, όπως και στα στις εθνικές κυβερνήσεις η δυνατότητα, εάν κάτι δεν γίνεται καλά, όπως όταν η κυβέρνηση δεν κάνει καλά τη δουλειά της πέφτει, έτσι πρέπει να γίνεται και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό λοιπόν σε γενικές γραμμές ε, συμφωνώ με τον συνάδελφο Ραγγέλ. Θα ήθελα να τον συγχαρώ και να του στήσω και συγγνώμη για την διακοπή. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω, ο κύριος Ράντζελ θέλει να συμπληρώσει τώρα ή να μιλήσει στο τέλο. Να, να συμπληρώσω, πέντε λεπτά μόνο. Γιατί και εγώ πρέπει να φύγω. Πρέπει να ολοκληρώσω την παρουσίασή μου. Λοιπόν... Όσον αφορά την νομοθετική πρωτοβουλία. Εδώ είναι σαφή τα πράγματα. Θα ήθελα όμως να αναφερθώ πολύ σύντομα και στις εξωτερικές σχέσεις. Προφανές είναι ότι η συνθήκη της Λισαβόνας έχει επιφέρει πολύ σημαντικές αλλαγές, ιδιαίτερα όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής στην περίπτωση, για παράδειγμα, της συμφωνίας SWIFT. Στην περίπτωση αυτή, τα άλλα θεσμικά όργανα, αλλά και οι εταίροι μας, από οι Πολιτείες, έχουν συνειδητοποιήσει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι μια υπολογίσιμη δύναμη, μια υπολογίσιμη εξουσία. Πώς να το πω. Υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες φυσικά, όμως σε γενικές γραμμές. Από τη στιγμή που εμείς καταψηφίσαμε τη συμφωνία SWIFT, η, ο Αμερικανός πρέσβης στη Λισαβόνα είχε τακτικές επαφές με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με ευρωβουλευτές και αυτό τι μας λέει, μας λέει ότι η Ουάσιγκτον πλέον έχει συνειδητοποιήσει ότι υπάρχουμε. Όταν ο Αμερικανός πρέσβης λοιπόν στη Λισαβόνα μέχρι τώρα μας καλούσε έτσι για τους τύπους και πλέον ζητεί επικοινωνία και συζήτηση για θέματα επί της ουσίας, αυτό δείχνει ότι έχει υπάρξει μια αλλαγή. Θέλουμε λοιπόν μηχανισμούς, θέλουμε διαδικασίες. Διαδικασίες ελέγχου ελέγχου των πληροφοριών στις διεθνείς συμφωνίες. Αυτό έγινε ήδη στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων για τη Συμφωνία Πλαίσιο. Είδαμε ότι πλέον υπάρχει επιθυμία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κάθεται και αυτό στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να μην απέχει. Και πιστεύω πως είναι πραγματικά κάτι που δεν, πρέπει, που δεν πρέπει να χάσουμε. Τα κοινοβούλια, βέβαια, δεν έχουν δημιουργηθεί για να κάνουν τέτοιες διαπραγματεύσεις. Αλλά εντάξει, εμείς έχουμε 700 ε, ευρωβουλευτές, έχουμε προσωπικό, αλλά σε γενικές γραμμές επίσης να πω ότι οι διαπραγματεύσεις πρέπει να γίνονται με διακριτικότητα και λαμβάνοντας πάντα υπόψη την εκτελεστική εξουσία που ασκούμε. Γι' αυτό δεν ε, αναφέρομαι μόνο και δεν κάνω μόνο απλές συστάσεις όσον αφορά τις ε, εξωτερικές ε, σχέσεις, αλλά εμβαθύνω στις σχέσεις μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Επίσης, αν κάνουμε τον απολογισμό των σχέσεων των θεσμικών οργάνων στα πλαίσια της ε, σύμβασης πλαισίου, τότε βλέπουμε ότι έχουν, έχει γίνει πρόοδος. Έχουν βελτιωθεί πολλοί σχέσεις Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κυρίως ε, εξαιτία της ε, σύμβάση πλαισίου. Και μπορούν να βελτιωθούν ακόμα περισσότερα πράγματα. Για παράδειγμα, οι πράξεις κατά εξουσιοδότηση ή οι ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προφορικές ή γραπτές, τα διάφορα μέτρα ή μελέτες που ζητούνται και διεξάγονται και οι νομοθετικές πρωτοβουλίες. Εδώ θα μπορούσαν να επέλθουν βελτιώσεις. Όμως αυτά που έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα, το Κοινοβούλιο δηλαδή να έχει περισσότερες Εξουσία είναι κάτι πάρα πολύ θετικό και να πω και κάτι άλλο, κάτι πολύ σημαντικό και πολύ αμφιλεγόμενο. Είναι σαφές ότι υπάρχουν ορισμένα θέματα τα οποία είναι σημαντικά, για παράδειγμα οι διμερείς σχέσεις Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και παραμένουν ανοιχτά ορισμένα θέματα τα οποία βρίσκουμε ξανά και στη συμφωνία πλαίσιο. Γι' αυτό ενδεχομένως χρειάζεται μια τρίμερη συμφωνία. Γι' αυτό πιστεύω πως θα ήταν καλό εάν το Κοινοβούλιο, η Κομισιόν και το Συμβούλιο κάθονταν μαζί για να δημιουργήσουν και να διαπραγματευτούν μια νέα τρίμερη συμφωνία για καλύτερη νομοθετική διαδικασία. Μόνο για ορισμένα ζητήματα της συμφωνίας πλαισίου. Αυτά θα μπορούσαμε να τα διαπραγματευτούμε και τα τρία θεσμικά όργανα και να οδηγηθούμε σε μια συμφωνία. Και αυτό θα σήμαινε, και αυτή είναι και η άποψή μου, ξέρω πως δεν θα συμφωνήσετε όλοι, θα σήμαινε λοιπόν ότι υπάρχουν σχέσεις Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Κομισιών, οι οποίες θα πρέπει να εξεταστούν διμερώς και όχι τριμερός. Αυτό το σημειώνω και στο τέλος της έκθεσης και εδώ στηρίζω τις τριμερείς συμφωνίες διότι είναι αναγκαίο και το Συμβούλιο να συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις έτσι ώστε να δημιουργείται μια πληρέστερη εικόνα και να οδηγούμαστε σε μια πληρέστερη συμφωνία. Όμως η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο πρέπει να δείξουν μεγάλη προσοχή για να μην χάσουν τις αρμοδιότητες που έχουν σε αυτές τις ε, τριμερείς ε, συμφωνίες και πρέπει να συζητηθούν εκεί μόνο αυτά τα σημεία που αφορούν και τα τρία θεσμικά όργανα. Ζητήματα συνταγματικής εφήσεως λοιπόν που αφορούν και τα τρία θεσμικά όργανα και από την άλλη μια διμερής ε, πλατφόρμα Συμβουλίου Κοινοβουλίου. Δύο λοιπόν είδη συμφωνίας και διαπραγμάτευσης και με αυτά ολοκληρώνω την παρέμβαση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκερέρο είναι ο πρώτος, πολλοί έχουν ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πάρα πολύ σύντομος, διότι ο ο ειδικό ε, σκιώδης εισηγητής ε, που έχει μακριά ιστορία εδώ είναι ο κύριος Λάιν. Εγώ θέλω να κάνω ένα σχόλιο μόνο για μία διάσταση που με ενδιαφέρει που είναι ο έλεγχος της Επιτροπής από το Κοινοβούλιο. Ο κύριος Ραγγέλ σε πολλές περιπτώσεις στην παρέμβασή του μίλησε για την ιδέα ότι δεν πρέπει να διευρύνουμε τις αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου, ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με τις αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου, ε, μιλώντας για το μεγάλο μεταπολεμικό συνταγματικό κίνημα που είναι ο εξορθολογισμένος συνταγματισμός, ε, κοινοβουλευτισμός που έχει προέλευση όχι στην γαλλική ημιπροεδρική στάση, αλλά στις αντιδράσεις για τις ε, προπολεμικές, μάλλον μέσοπολεμικές ε, ε, πολιτικές αστάθειες, κυρίως στη Βαϊμάρη. Σαν αποτέλεσμα της αστάθειας αυτής είχε προκύψει ότι ε, οι κοινοβουλευτικές δομές μετατρέπονταν σταδιακά σε κυβερνώσεις βουλές, με αποτέλεσμα στην πλειοψηφία των περιπτώσεων περιπτώσεων η νομοποίηση των κυβερνήσεων εν τέλει να είναι μια άμεση νομοποίηση από πλευρά πολιτών που ψηφίζουν προγράμματα και υποψήφια. Οπότε ολόκληρη η δυναμική του δεύτερου τμήματος του 20ου αιώνα ήταν μια δυναμική ενίσχυση των κυβερνήσεων και αποδυνάμωση των κοινοβουλίων σαν αντίδραση στην προγενέστερη αυτή τάση. Με την πάροδο του χρόνου εμφανίστηκαν τα προβλήματα που θέτει ο εξορθολογισμένος κοινοβουλευτισμός, δηλαδή η πραγματική και ουσιαστική δυσκολία ελέγχου των κυβερνήσεων. Όχι υποκατάσταση των κυβερνήσεων στην εκτελεστική εξουσία, αλλά στην, ε, στον έλεγχο του τι κάνουν. Θα ήταν κάπως περίεργο, αυτό που, θα ήταν, περί, που ήταν περίεργο μάλλον, είναι ότι ο ξεδοθολογισμένος κοινοβουλευτισμός είναι κάτι που ενδιαφέρει ιδίω τις κυβερνήσεις. Και οι κυβερνήσεις ήταν αυτές οι οποίες ε, πίεσαν προς την τάση αυτή και άρα είναι κάπως περίεργο ένα κοινοβούλιο να παροτρύνει την αποδυνάμωσή του, την ίδια αποδυνάμωσή του. Αυτό είναι συζητήσιμο. Ξέρω ότι είναι συζητήσιμο, διότι ο καθηγητής κ. Ζαντζέλ τόνισε, και εγώ συμφωνώ μαζί του, ότι δεν πρέπει να υποκαταστήσουμε την κυβέρνηση από την αρμοδιότητά της ως, ε, ως όργανο εκτέλεσης των αποφάσεων, αλλά γι' αυτό το λόγο πρέπει να αυξήσει να αυξήσουμε τον έλεγχο του Κοινοβουλίου στις εκτελεστικές δομές και αυτό σημαίνει να μην αποποιηθούμε την δυνατότητα απέτηση πολιτικής ευθύνης από την Επιτροπή. Είναι γεγονός ότι αυτό μπορούμε να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει κάτι τέτοιο, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι καλό σύστημα να λέμε ότι καταρχήν ε, δεν θέλουμε να απαιτήσουμε πολιτική ευθύνη από έναν επίτροπο συγκεκριμένα μεταξύ πραγμάτων που τίθενται ή να συζητήσουμε τις πλειοψηφίες, τη διαδικασία, ναι, αλλά το να αποποιηθούμε αφεαυτού μια τέτοια δυνατότητα το θεωρώ λάθος. Αύξηση ελέγχου σημαίνει και λογοδοσία. Εμείς έχουμε πολλά θέματα επιτάπητος, φερπίν τον έλεγχο από το Κοινοβούλιο στην ε, λειτουργία της Τρόικα ή την απέτηση, στην απέτηση, της, την απέτηση να απαντα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε ερωτήσει του, του Κοινοβουλίου. Ο Ρομπέρτο θα σα μιλήσει για τα ζητήματα που τίθενται και του μηχανισμού που ανακύπτουν από την οικονομική διακυβέρνηση, το μηχανισμό σταθερότητα. Το τι θα γίνει στο μέλλον, α πούμε, όταν κάποιε από τι συνθήκε που εγκρίθηκαν με διακυβερνητικό τρόπο αρχίσει να, αρχίσουν να εισέρχονται στην ε, νομοθεσία της Ένωσης, δηλαδή της συνθήκης. Τέλος πάντων, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, να πω απλά ότι με ανησυχεί η δυνατότητα ως κοινοβούλιο ε, πάμε στο να αποδυναμώσουμε τη θέση του κοινοβουλίου. Δεν κάνω πρόταση υπέρ του να κυβερνά την Ευρωπαϊκή Ένωση το Κοινοβούλιο. Εγώ συμφωνώ με την ιδέα ότι άλλος κυβερνά, άλλος νομοθετεί αλλά στην περίπτωση αυτή πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα αυστηροί και φιλόδοξοι στη διαμόρφωση μηχανισμών υπευθυνότητα στενή ενία και ελέγχου υπό την έννοια της λογοδοσίας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντάφ τώρα. Um, uh, thank... Κύριε Πρόεδρε, Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω θερμά τον Πάλο Ρανζέλ και για την έκθεσή του, αλλά και για την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα γνωμοδότηση που έχει συντάξει. Νομίζω ότι εδώ μπορούμε να διαπιστώσουμε κάποιες πολύ σημαντικές ιδέες για μια μελλοντική συντακτική συνέλευση και στο τέλος της ε, έκθεσης θα μπορούσαμε ίσως πιο συγκεκριμένα να αναφέρουμε εμείς ως Επιτροπή συγκεκριμένα τι θα θέλαμε να συμπεριληφθεί ε, στην ε, ατζέντα, στην μέση διάταξη της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, στη συντακτική συνέλευση. Κάτι αντίστοιχο δηλαδή με την προσέγγιση που ακολουθήσαμε στην έκθεση Γκουαλτιέρη Τρασκόφσκι. Νομίζω ότι αυτό το στυλ, ε, ο τύπος που είχαμε βρει είναι καλός και θα μπορούσαμε να τον αντιγράψουμε και στην προκειμένη περίπτωση. Δεύτερον, συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα ότι αυτό το οποίο προσπαθούμε να οικοδομήσουμε, δηλαδή μια κοινοβουλευτική και όχι μια προεδρική Ευρώπη, είναι ε, σωστός στόχος, αλλά θα πρέπει να το κάνουμε με ένα ομόσπονδο ή αναδιόμενο αν θέλετε ε, ομόσπονδο σύστημα και είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη μας το Ινδικό και ε, Καναδικό παράδειγμα. Ανέφερε τα σχετικά ο εισηγητής, δηλαδή βασίστηκαν στην Βρετανική εμπειρία. Ομόσπονδα συστήματα κατ' ουσίαν είναι δεν μπορούμε να είμαστε πάρα πολύ κατηγορηματικοί και απόλυτοι αυτή τη στιγμή ως προς το είδος της Προεδρίας θα προκύψει. Νομίζω ότι άμεσα, άμεσα αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο προέχει είναι αυτή τη διάχυτη εκτελεστική αρχή, την κατακαιρματισμένη, την αδιαφανή, να την συγκεντρώσουμε κατά κάποιο τρόπο. Να τη συγκεντρώσουμε στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και βέβαια αυτό σίγουρα δυνητικά δίνει τεράστια δύναμη στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ προσωπικά ελπίζω αυτό το νέο πείραμα το οποίο θέλουμε να εφαρμόσουμε, δηλαδή την εκλογή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ελπίζω λοιπόν αυτό να, να δώσει στον Πρόεδρο αυτό ε, μία διπλή νομιμοποίηση, δηλαδή νομιμοποίηση και από το Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο. Οπότε θα μπορεί το άτομο αυτό να ασκεί μεγαλύτερη επιρροή στη διαμόρφωση ε, και τη σύνθεση του σώματος ε, των επιτρόπων και θα έχει μεταξύ άλλων και την ε, εξουσία να απορρίπτει υποψηφίους που ενδεχομένως δεν συμφωνεί να είναι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 7 Ιουλίου θα έρθει και ο υποψήφιος, θα έρθουν μάλλον οι υποψήφοι για τη θέση του Πρόεδρου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Θα γίνει στο, με το σχηματισμό της διάσκεψης των Προέδρων. Θα είναι καλύτερη, πιστεύω, αυτή η συνεδρίαση, αν γίνει κάπως ευρύτερα από ό,τι γινόταν μέχρι τώρα και αν μπορεί να συγκριθεί με τις ακροάσεις που πολύ επιτυχημένα μέχρι τώρα έχουμε διεξαγάγει για τα μεμονωμένα μέλη των επιτρόπων. Τις επιτρόπεις, τους επιτρόπους τέλος πάντων. Τι, το φθινόπωρο διεξάγονται οι ακροάσεις αυτές. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους μεμονωμένους επιτρόπους ε, και την εκλογή τους, τα χαρτοφυλάκια τους, αυτά θα πρέπει να τα δούμε, να εμβαθύνουμε. Δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει το κοινοβούλιο. να έχει κάποιες ε, δυνατότητες ε, λογοκρισία, μομφής μάλλον απέναντι στους επιτρόπους Έχουμε και κάποια υπόθεση, κάποια παρελθόν στη Βρετανική ε, ιστορία. Αλλά στο Westminster ε, το σύστημα ε, επιτρέπει μεγάλο έλεγχο στην εκτελεστική εξουσία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη σχέση μεταξύ Κοινοβουλίου και Κομισιών, ξέρουμε την προβλέπει η της Λισαβόνας. Ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε με τη δεύτερη βουλή, κατά κάποιο τρόπο, ε, το νομοθετικό Συμβουλίο Υπουργών. Την αποτελεσματικότητα των συναντέλφων στο Συμβούλιο. Και βέβαια αυτό θα μας οδηγήσει και σε μια ακόμη σκέψη ε, του Συμβουλίου της Ένωσης. Ποιος είναι ο ρόλος, ποιες είναι οι σχέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ενεκρίθη πρόσφατα έκθεση Λαμασούρ επί του θέματος. Βέβαια, προσωπική μου άποψη είναι ότι θα μπορούσε να πάει πιο μακριά η έκθεση. Θα μπορούσε δηλαδή να προτείνει ε, κάποιες επιλογές, κάποιες συναλλακτικές για τη μεταρρύθμιση αυτού του οργάνου λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της συνθήκης της Λισαβόνας. Επομένως, νομίζω είναι μια εξαιρετική αφετηρία ε, για να μπορέσουμε να καταθέσουμε πολλές ε, τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ο κ. Λάινεν έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σε δύο μέρες ήρθα. Ήρθα δύο φορές σε δύο μέρες μάλλον. Χθες μίλησα, αλλά και το θέμα αυτό με απασχολεί πάρα πολύ καιρό. Με απασχολεί από την προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Ρανζέλ για την ε, πολύ σημαντική έκθεση. Να πω ότι στην ε, τελευταία συνεδρίαση, σε 7 Μαΐου του 2009, την προηγούμενη νομοθετική περίοδο, την προηγούμενη θητεία δηλαδή, είχε υποβληθεί στην Ολομέλεια μία έκθεση για τις αρμοδιότητες και τις ε, εξουσίες ε, του Κοινοβουλίου μετά από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Εισηγητής ήταν ο υποφαινόμενος. Μπορείτε όσοι έχετε έρθει μετά από μένα να δείτε την έκθεση, να τη διαβάσετε, είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες και σα το προτείνω αυτό γιατί τότε κοιτάξαμε πάρα πολύ αναλυτικά τη συνθήκη της Λισαβόνας και τι αυτή επιφέρει. του νέους στόχους, οριζόντιες ε, ε, νέα νομική βάση, συναπόφαση νέε δημοσιονομικέ αρμοδιότητες, νέα διαδικασία ψηφοφορίας, νέες ε, αρμοδι... και εποπτικές αρμοδιότητες, δικαίωμα πρωτοβουλίας κλπ. κλπ. Επομένως, μετά από την ε, συνθήκη της Λισαβόνας αποκτήσαμε πάρα πολλές εξουσίες, ε, σημαντικές εξουσίες και είναι πάρα πολύ σημαντικό θεωρώ στο τέλος της, ε, νομοθετικής θητείας, της κοινοβουλευτικής θητείας να κάνουμε τον απολογισμό μας και να δούμε τι λειτουργεί και τι όχι και τι όχι τόσο καλά. Εάν πάρουμε στα σοβαρά τον τίτλο της έκθεσης, εφαρμογή δηλαδή της θήκης της Λισαβόνας με βάση τα δικαιώματά μας, θα συνειδητοποιήσουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ακριβείς προγνώσεις ε, για το μέλλον. Έχουμε ήδη κάνει πάρα πολλές σχετικές εκθέσεις. Η έκθεση Tyson, για παράδειγμα, ήταν μια έκθεση η οποία ασχολήθηκε πάρα πολύ με το υπόβαθρο και το χαρακτήρα που κινδυνεύει να χαθεί. Ασχοληθήκαμε λοιπόν με την ενίσχυση του δημοκρατικού ελέγχου και είδαμε πού ε, όντω ενισχύθηκε, πού όχι, ποιοι κίνδυνοι υπάρχουν. Και εμεί ε, ε, κάναμε μία έκκληση για την όσο το δυνατόν γρηγορότερη εφαρμογή. Τώρα, όσον αφορά την ε, νομοθεσία, η συνθήκη της Λισαβόνας αναφέρεται στη συνήθη νομοθετική διαδικασία δηλαδή συναπόφαση και εδώ πρέπει να κοιτάξουμε τα σημεία στα οποία η διαδικασία συναπόφασης δεν λειτουργήσε καλά και που φταίμε εμείς. Το είπαμε ήδη πολύ συχνά, το έχουμε πει στο παρελθόν ότι υπάρχουν ορισμένες τάσεις που έχουν ε, ε, παρατηρηθεί. Να παρακάμπτεται η συνήθιση νομοθετική διαδικασία μέσω διαδικασιών του Συμβουλίου, για παράδειγμα, μέσω πράξεων οι οποίες μας παρακάμπτουν. Και αυτά πρέπει να τα κατονομάσουμε. Μετά υπήρξε μια γνωμοδότηση της Επιτροπής ΙΝΤΑ, ΛΥΜΠΕ και Γιούρι, αυτών των τριών επιτροπών. Θα ήθελα πάρα πολύ να είχαν γνωμοδοτήσει και οι Επιτροπές Νομισματικών Οικονομικών Υποθέσεων και η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων διότι ιδιαίτερα όσον αφορά τη δημοσιονομική, οικονομική πολιτική, την οικονομική άμυνας και ασφάλειας και, τον, ε, και εξαιτία του παλαιότερου τρίτου πυλώνα έχουν δημιουργηθεί γκρίζε ζώνε, Έχουμε μεν αποκτήσει νέα δικαιώματα, όμω μετά τις ε, επικαλύψεις ε, αρμοδιοτήτων ε, ελοχεύει ο κίνδυνο να αποκλειστεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την νομοθετική διαδικασία. Ε, τομείς που λειτουργούν καλά μετά τη συνθήκη τη Λισαβόνα είναι η κοινή αλληλευτική πολιτική και εδώ βλέπουμε ότι η, συνήθ, ότι η διαδικασία συναπόφαση έχει λειτουργήσει πάρα πολύ καλά και έχει επιφέρει πλέον εκτήματα. Τώρα, από το, τώρα το 2014. Το κύριο σημείο που θα μας απασχολήσει είναι η εκλογή του Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η νέα αρμοδιότητα που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκλέξει τον Πρόεδρο και όχι απλά έτσι να ε, λειτουργεί ήδη και απλά να εγκρίνει. Υπάρχουν ε, σαφείς προδιαγραφές ε, πλέον του Κοινοβουλίου που ε, σκεγγραφούν το τι θέλουμε από έναν πρόεδρο της Επιτροπής και υπάρχει και ένας νέος μηχανισμός σαφώς καθορισμένος που προβλέπει την ε, διαδικασία και τις λεπτομέρειες αυτής. Έχουν ήδη συζητηθεί αυτά τα θέματα. Τώρα υπάρχουν πλέον ε, νέα δικαιώματα συναπόφασης, ορισμός για παράδειγμα προσώπων και εδώ έχουμε διατυπώσει τις θέσεις και τις επιθυμίες μας. Ο συνάδελφος Ραντζέλ επίσης πολύ σωστά είπε ότι δύσκολα μπορούμε να λάβουμε σωστή απόφαση αν δεν έχουμε πληροφορηθεί επαρκώς. Και εδώ υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες ε, είναι εκεί, η πράσινη χάρτα, δια, διοργανικές συμφωνίες για την νομοθεσία και Αυτές ε, τις ε, δυνατότητες που έχουμε πρέπει να τις αναλύσουμε διεξοδικά για να δούμε πώς μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε. Τώρα, πράξεις κατά εξουσιοδότηση είναι πάρα πολύ σημαντικές. Έχουμε ένα νέο σύστημα πλέον με τη συνθήκη της Λισαβόνας όπου οι... πολλαπλασιάστηκαν οι αρμοδιότητές μας και οι εξουσίες μας. Στην τελευταία θητεία είπαμε ότι υπάρχουν 300 νόμοι και 300.000 ε, πράξεις κατά εξουσιοδότηση. Πιο πολλές δηλαδή από ότι νόμους. Και στις πράξεις ε, κατά εξουσιοδότηση κρύβονται πάρα πολλές λεπτομέρειες και υπάρχει αυτός ο ένας ε, πόλεμος ανάμεσα σε εκτελεστικές πράξεις και πράξεις κατά εξουσιοδότηση. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να τονιστεί και πολύ σωστά γίνεται στην έκθεση. Επίσης, να πω ότι ένα δικαίωμα το οποίο αποκτήσαμε και δεν έχουμε πάρει στα σοβαρά μέχρι τώρα είναι το δικαίωμα της πρωτοβουλίας για αλλαγή των συνθήκων. Έχουμε ε, πολλούς τομείς όπου διατυπώθηκαν πολλές νέες επιθυμίες και πιστεύω πως αυτή η έκθεση θα πρέπει να συμπεριλάβει ε, και κάποιο στοιχείο για ενίσχυση του δημοκρατικού ελέγχου και ενίσχυση της διαπραγματευτικής δυνατότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να γίνουν όλα αυτά χρειάζονται βελτιώσεις τις οποίες η, η συνθήκη της Ελισαβόνας δεν προβλέπει τόσο έντονα. Αυτό λοιπόν το δικαίωμα πρωτοβουλίας που αποκτήσαμε είναι κάτι το οποίο δεν χρησιμοποιήσαμε στο έπακρο σε αυτήν την κοινοβουλευτική θητεία και πιστεύω πως εντάξει, αυτή η έκθεση δεν θα το ε, αναπτύξει όσο θα έπρεπε. Αυτά από εμένα, κύριε συνάδελφε Ράγκελ, χαίρομαι πάρα πολύ για την έκθεση. Ελπίζω σε μια πολύ καλή συνεργασία θα σας κατακλείσω με τροπολογίες και να πω ότι η εφαρμογή της ε, συνθήκης ε, της Λισαβόνας, ε, η θέση ισχύ μάλλον της, της συνθήκης της Λισαβόνας μας έφερε νέες αρμοδιότητες τις οποίες έχουμε καλωσορίσει. Ένα πράγμα επίσης με βρίσκει πάρα πολύ σύμφωνο, ένας κατάλογος απαιτήσεων για τον ε, εκλεγέντα πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2014. Χρειαζόμαστε λοιπόν έναν τέτοιο κατάλογο. Αλλά χρειαζόμαστε, χρειάζεται να δούμε και το Συμβούλιο και το τι αυτό πρέπει να αλλάξει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα πάντα καλύπτει η έκθεση Ρανζέλ ξεκίνησε από τον Μοντεσκέ για την διάκριση των εξουσιών μέχρι σήμερα. Εγώ θα συμφωνήσω με τον Άντριου Νταφ. Το μέλλον της Ευρώπης είναι κοινοβουλευτικό, όχι προεδρικό. Ούτε καν ο ημιπροεδρισμός που αναδεικνύεται, παρότι κανείς δεν το λέει έτσι, είναι κάτι που πρέπει να παρακολουθήσουμε προσεκτικά. Επίσης, είναι σημαντικό κάπου στην έκθεση να επανεπιβεβαιωθεί η λαϊκή κυριαρχία που υπάρχει, που εκπροσωπείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κυριαρχία που από ό,τι φαίνεται δεν το γνωρίζει η πλειοψηφία του κόσμου. Άλλο το θέμα αυτό όμως τόσο. Σε ό,τι αφορά τα προεδρικά συστήματα, Η επίσκεψη που κάναμε πριν από λίγες εβδομάδες στην, ε, στη Ουάσιγκτον με οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι ναι, μεν είναι προεδρικό το σύστημα στη ΣΥΠΑ, αλλά μοιάζει πολύ περισσότερο με κοινοβουλευτικό από ό,τι ε, φαίνεται. Διότι ο πρόεδρο για να πετύχει κάτι, ό,τι και να είναι, πρέπει να έχει την υποστήριξη της, ε, του, των νομοθετικών σωμάτων. Που δεν το κάνει αυτή τη στιγμή. Οι υπερβολικοί έλεγχοι και ισορροπίες οδηγούν σε διέξοδα. Πρέπει λοιπόν να έχουμε επίγνωση ότι όταν διαμορφώνουμε, διαμορφώνουμε πιο σωστά το σύστημα, το θέμα των ελέγχων και ισορροπιών θα πρέπει να το σκεφτόμαστε προσεκτικά και να το διορθώνουμε όπου χρειάζεται. Στο πλαίσιο αυτό, και νομίζω ότι η έκθεση αυτό λέει, αλλά μπορεί να το πάω προς μια κατεύθυνση που δεν θέλει ο Παύλο Ρανζέλ, είναι ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε πω η Επιτροπή ασκεί εξουσίε. Φερρυπίν, αδιαμφισβήτητα το δικαίωμα τη νομοθετική πρωτοβουλία είναι άσκηση εξουσία. Αυτό τι σημαίνει ότι η Επιτροπή κατά συνέπεια έχει κάποια, κάποιο κομμάτι κυριαρχία από τα κράτη-μέλη. Και ναι, τι, ποιο επίπεδο, πώ εμπλέκεται το, το Συμβούλιο, και μια ερώτηση που θα μπορούσα να θέσω είναι στο πλαίσιο της ε, μορφής επιμέρους επιτρόπων μήπως ήταν λογικό να εκλέγει το κάθε επίτροπος απευθείας από κάθε κρατός Έτσι αλλάζει και η ισορροπία. Ιδέα είναι. Μετά, είναι γεγονός ότι η διακυβέρνηση είναι τεχνική. Γίνεται όλο και περισσότερο τεχνική. Που σημαίνει ότι όταν έχουμε 28 κράτη η τεχνικότητα μετα... ενισχύεται. Και το πολιτικό στοιχείο των δράσεων της Επιτροπής δεν γίνεται αποδεκτό. Θα έπρεπε να ξέρουμε επίσης ότι η αύξηση της νομοθετικοποίηση της πολιτικής, δηλαδή το να πολιτική μέσω διοικητικών και νομοθετικών πράξεων, ε, δημιουργεί κινδύνους. Από την άλλη μεριά, οι ασυμμετρίες εξουσίας νομίζω ότι ουδέποτε μπορούν να παραμεριστούν, πάντα θα υπάρχουν δεν πρέπει να μας ανησυχούν αυτές, αλλά οι μηχανισμοί. Γιατί εγώ πιστεύω ότι η διαφάνεια και η λογοδοσία είναι ζωτική σημασίας, η διαθεσιμότητα πληροφοριών επίσης, η πλήρης ενημέρωση και το feedback και η αμοιβαιότητα στην παροχή πληροφοριών. Μια άλλη άποψη μια, κάποια σκέψη ακόμα. Το επόμενο κοινοβούλιο και φαντάζομαι θα είναι διαφορετικό από το τωρινό. Και δεν είμαι ο μόνος που το φαντάζεται. Υπάρχουν ε, οι γενικές αρχές βέβαια της διαιώνισης του κοινοβουλίου, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το context όταν ε, νομοθετούμε. Άρα πρέπει να έχουμε υπόψη και το βραχυπρόθεσμο. Τι κοινοβούλιο δηλαδή θα δώσουν οι ευρωεκλογέ του Μαΐου. Ευχαριστώ κύριε Σέπλιν, ο κύριος Χέφνερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ και τον Παούλιο Ραγγέλ για το σχέδιο έκθεσης και για, την, ε, για τις ιδέες του. Πιστεύω πως ε, ασχολείται με πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα, την εφαρμογή και τις πρακτικές εμπειρίες που έχουμε αποκομίσει από την ε, η συνθήκη της Λισαβόνας, ιδιαίτερα όσον αφορά τις σχέσεις Κοινοβουλίου και Κομισιών και τον απολογισμό που κάνει από αυτό. Θα ήθελα να πω καταρχάς ότι η έκθεση αυτή χρειάζεται να εξεταστεί λεπτομερώς πρωτού υποβάλλουμε πρωτοβουλίες και αυτό το λέω γιατί ε, πήρα μόλις χθε το σχέδιο έκθεσης και το διάβασα με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όμως σε γενικές γραμμές πιστεύω πως ε, η αναλογία χρόνου που έχουμε να διαβάσουμε μια έκθεση και εμβάθυνσης που μπορούμε να κάνουμε δεν φτάνει. Πιστεύω πως έχουμε πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα να συζητήσουμε και να ασχοληθούμε και χρειάζεται μήνες προετοιμασίας ε, και όχι απλά λίγες μέρες. Γι' αυτό λοιπόν ε, θα ήθελα πρωτού συζητήσω επί του περιεχομένου να έχω τον χρόνο μια τέτοια έκθεση έχει, που ανακοινώνεται μήνες πριν και φτάνει στα χέρια μας ώρες πριν, δεν μπορεί να απολαύσει μια καλή συζήτηση στην Επιτροπή. Όπως και η έκθεση Λαμασούρ, για παράδειγμα. Πιστεύω πως εδώ πέρα υπάρχουν ελλείψεις στην διαδικασία. Αυτά ως προς την μέθοδο και το χρονοδιάγραμμα. Τώρα όμως, ε, για το περιεχόμενο, να πω ότι η μεγάλη γραμμή που υπάρχει εδώ, για εμένα και για την ομάδα μου, όσον αφορά τις προτάσεις και διαπιστώσεις του Παόλιο Ραντζέλ είναι η διάκριση των εξουσιών, η ενίσχυση της διάκρισης των εξουσιών και της ε, δημοκρατίας. Εδώ πέρα συμφωνούμε και υποστηρίζουμε τον Πάουλο Ραντζέλ απόλυτα και να πω σύντομα ότι καταρχάς η μελλοντική, η μελλοντική επίτροπη θα μπορούν πλέον να προέρχονται και από τις τάξεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα έπρεπε ίσως να προέρχονται και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό το θεωρούμε ένα πολύ ωφέλιμο και σημαντικό βήμα προς τα μπροστά. Ο, τώρα, εντάξει, η διατύπωση της έκθεσης δεν με βρίσκει και απόλυτα σύμφωνο. Υπάρχουν, για παράδειγμα, ορισμένες διατυπώσεις όπως το newly elected πρόσφατα εκλεγμένος. Ε, εντάξει, δεν είναι απαραίτητο να είναι λοιπόν πρόσφατα εκλεγμένοι. Χρειάζεται να είναι εκλεγμένα μέλη. Μπορούν να είναι πιο παλιά, να έχουν περισσότερη πείρα. Επίσης, ακόμα περισσότερο σημαντικό μου φαίνεται ότι υπάρχει η πρόταση για τρεις προτάσεις για τον πρόεδρο της Επιτροπής και όχι για έναν. Εδώ, εδώ θα έχουμε πλέον μεγαλύτερο περιθώριο ελιγμών, μεγαλύτερη ελευθερία και πιστεύω πως αυτή την, ε, αυτή την εποχή έτσι όπως είναι η, κατάσταση είναι, μας υπαγορεύει σχεδόν μας υπαγορεύουν οι εθνικές κυβερνήσεις ε, τον υποψήφιο, δεν μας δίνουν το περιθώριο της ε, επιλογής και πιστεύω πως χρειάζεται να διασφαλίσουμε την δυνατότητα επιλογής, της περισσότερες επιλογές Αυτό οδηγεί σε περισσότερη δημοκρατία και θα οδηγήσει επίσης και σε αύξηση της ποιότητας, διότι αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη έχουμε προβλήματα και δεν πρέπει να δεχόμαστε τις δεύτερες και τρίτες επιλογές όπως ε, είναι μέχρι τώρα. Τότε θα έχουμε την δυνατότητα να επιλέξουμε πραγματικά τον καταλληλότερο άνθρωπο για την σωστή θέση. Και αυτό θα γίνει με την αύξηση των υποψηφίων από έναν σε τρεις. Τώρα, έχω ορισμένες αμφιβολίες για το θέμα της περιτροπής ε, αλλαγής των χαρτοφυλακίων των επιτρόπων. Πιστεύω πως εδώ προσπαθούμε να τετραγωνίσουμε τον κύκλο. Από τη μία να μειώσουμε τον αριθμό των επιτρόπων, να μειώσουμε την ε, έκταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά να μην χάσουμε και κανέναν επίτροπο, να παραμείνουν οι ίδιοι. Και αυτή η ιδέα των ε, επιτρόπων ανευχαρτοφυλακίου μου ε, ξυπνά ανησυχίε, διότι τι θα κάνει ένας επίτροπος πέντε χρόνια. Στη Μεγάλη Βρετανία τους θεωρούν αδέσποτους και απρόβλεπτους. Κα, κάποια αρμοδιότητα πρέπει να υπάρχει. Δεν μπορεί ένας επίτροπος να μην έχει αρμοδιότητες. Πρέπει να αναπτύξει το δικό του προφίλ, να κάνει το δικό του έργο. Δεν μπορούμε δηλαδή να έχουμε τη μισή επιτροπή με χαρτοφυλάκιο και την άλλη μισή λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Μου φαίνεται κάπως ύποπτη λοιπόν αυτή η πρόταση. Έπειτα, όσον αφορά την άμεση εκλογή του Προεδρού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτή είναι μία πρόταση η οποία Φαίνεται πως ε, επιφέρει περισσότερη δημοκρατία, όμως στην πραγματικότητα καταφέρνει το αντίθετο αυτό το προεδρικό σύστημα. Πιστεύω πως δεν έχουμε σκεφτεί μέχρι τέλους όλες τις επιπτώσεις ενός τέτοιου προεδρικού συστήματος. Και να σας υπενθυμίσω και την ακρόση που έχουμε προγραμματίσει για το 2014 για το πρώτο μισό του 2014, όπου τότε θα συζητήσουμε διεξοδικά το ζήτημα αυτό θα είναι πιστεύω μια πάρα πολύ σημαντική και χρήσιμη συζήτηση και εγώ τουλάχιστον θεωρώ απαραίτητο ένα σύστημα κοινοβουλευτικής αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, ε, κοινοβουλευτικό χαρακτήρα, ενίσχυση του κοινοβουλευτικού χαρακτήρα. Επίσης, σημαντικό θεωρώ το σημείο 11 και 20. Εκεί όπου αναφέρεται δηλαδή ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα μπορεί πλέον να αγνοεί τις συστάσεις και τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και όπως είπε και ο Έλμαρ Μπρόκ πιο πριν, αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να συζητήσουμε με τον νέο υποψήφιο για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το δικαίωμα της συναπόφασης και πρέπει η θέση του Προέδρου της Επιτροπής να είναι όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητη. Ένα κοινοβούλιο χωρίς λειτουργικά, απτά δικαιώματα νομοθετικά μου φαίνεται πως είναι πολύ αδύναμο. Δεν πρέπει να περιοριστούμε στην αντίδραση, πρέπει να αναλάβουμε και δράση. Και να ζητούμε λογοδοσία, να ζητούμε αιτιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε περίπτωση που αρνείται να, να λάβει υπόψη την άποψή μας. Διότι αυτό το θεωρώ απαράδεκτο. Τώρα, ε, όσον αφορά το πρόβλημα των ε, πράξεων κατά και των εκτελεστικών πράξεων, εδώ με ανησυχεί κάπως η διατύπωση, διότι ε, πιστεύω πως δεν θα αλλάξει ουσιαστικά την υφιστάμενη κατάσταση. Και πρέπει να δούμε πώς θα αλλάξει αυτό, τι μπορούμε να κάνουμε στον τομέα αυτό. Σε γενικές γραμμές όμως πιστεύω πως θα αλλαξει αυτο τι μπορουμε να κανουμε στον τομεα αυτο σε γενικε γραμμες ομως πιστευω πως ειναι μια πάρα πολύ καλή βάση το αυτό το σχέδιο έκθεσης για περαιτέρω συζήτηση και επεξεργασία στην Επιτροπή και ε, θα έχουμε, είμαι σίγουρο, τη δυνατότητα στην ε, ομάδα των σκιωδών εισηγητών και στην Επιτροπή να λάβουμε υπόψη όλε τι προτάσει και να δημιουργήσουμε κάτι πραγματικά αξιόλογο. Σα ευχαριστώ πολύ. Thank you. I, Ο κύριος Μπρόντς. Σήμερα το πρωί το είδα. Αλλά θα σταθώ μόνο σε ένα τμήμα και αυτό θα χαροποιήσει τους διερμηνείς φαντάζομαι. Στην παράγραφο Α, πρόταση 3 της έκθεσης. Την έμεση εκλογή του Πρόεδρου της Επιτροπής. Η άποψη των ψηφοφόρων θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στην επιλογή του Πρόεδρου. Αν όλοι οι περισσότεροι ε, ψηφοφόροι ψηφίσουν, ψηφίζουν ευρωπαϊκά και όχι εθνικά πολιτικά κόμματα που μπορεί να είναι ή να μην είναι μέρη ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και εφόσον το έκανα με βάση το κριτήριο του ορισμού ε, του συγκεκριμένου υποψηφίου από τα κόμματα, τότε όντως ο ψηφοφόρος κάνει επιλογή. Αν ωστόσο οι ψηφοφόροι συνεχίζουν να ψηφίζουν εθνικά πολιτικά κόμματα, είτε είναι είτε δεν είναι μέρη πολιτικών κομμάτων, ή ψηφίσουν για πολιτικά κόμματα μόνο διότι αυτό το κόμμα θέλουν σε εθνικό επίπεδο, δεν νομίζω ότι μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζεται η άποψη του ψηφοφόρου στην, στον, επί, στον πρόεδρο τη Επιτροπή. Τα κριτήρια δεν μπορεί να, να υποχρεωθούν να ακολουθήσουν συγκεκριμένα κριτήρια, όπω μπορεί να υποχρεωθούν να ψηφίσουν με συγκεκριμένο τρόπο. Κατά συνέπεια, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι οι ψηφοφόροι που ψηφίζουν ένα συγκεκριμένο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα, στο οποίο παράδειγμα είναι μέλη οι φιλελεύθεροι, υπερψηφίζουν το κόμμα αυτό λόγω του υποψηφίου της Επιτροπής μπορεί να ψηφίζουν το κόμμα αυτό γιατί είναι κομμάτι, γιατί κομμάτι του κόμματος αυτού είναι φιλελεύθεροι. Οι ψηφοφόροι στη Βρετανία, δεν μπορώ να μιλήσω για όλες τις χώρες της Ένωσης, κατά πάσα πιθανότητα ουδέποτε έχουν ακούσει για ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Πολλοί δεν έχουν ακούσει καν για επιτροπή ή για πρόεδρο της επιτροπής. Και αυτό είναι και κάποιο, το, πιο, το χειρότερο όλων δεν είναι ότι κάποιοι μπορεί να έχουν ακούσει καν για ευρωβουλευτές. Δεν λέω ότι αυτό είναι καλό. Καλό θα ήταν να είναι ενημερωμένοι. Αλλά το επίπεδο ενημέρωσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση στα κράτη-μέλη φοβάμαι ότι είναι μάλλον ε, χαμηλό. Θα απαιτηθούν χρόνια επανεκπαίδευσης, ό,τι είναι ο όρος αυτό, για να τους εξηγήσουμε τι σημαίνουν οι όροι αυτοί και να τους πείσουμε να ψηφίσουν βάση συγκεκριμένου υποψήφιου για την Προεδρία της Επιτροπής. Αυτά ήθελα να πω μόνο. Ευχαριστούμε. Κύριε Μπρόντς, ο κύριος Γκουαλτιέρη. Ακόμα και εγώ θα είμαι πολύ σύντομος, πρόεδρε, γιατί οι συνάδελφοι Γκερέο και Νταφ τάπανε και παρουσίασαν τη θέση της ομάδας για την έκθεση που περιλαμβάνει πολλά ενδιαφέροντα σημεία. Με άλλα συμφωνούμε, με άλλα πρέπει να τα δούμε πιο προσεκτικά και εκεί θα υποβάλουμε το υπολογίσμα Θα σταθώ σε ένα ζήτημα μόνο. τον ρόλο του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της οικονομικής και νομισματικής πολιτικής της Ένωσης. Προφανώς ε, εκτεταμένο θέμα που καλύπτει και η έκθεση που έχω κάνει με τον κύριο Τραζακόφσκι αλλά και δεν πιστεύω ότι πρέπει να επανεισαχθεί στην έκθεση αυτή όπως έχει, αλλά υπάρχει ένα ζήτημα που νομίζω ότι θα έπρεπε για να έχει συνοχή να αποτελεί κομμάτι της έκθεσης ε, Ραγγέλ. Και ξεκινάω με μια διαπίστωση ότι είναι αδιαμφισβήτητο ότι τη στιγμή που μέσω μιας σειράς νέων νόμων και μέσω μιας ενίσχυσης του ρόλου τη ε, υποδηλούμενη πολιτική πίεση που συνδέεται με το γεγονό ότι και άλλοι οργανισμοί όπως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας είναι ε, δομέ που παίρνουν αποφάσεις καθοριστικέ για κάποιες χώρες. Από τη στιγμή που αρχίζουν να λειτουργούν αυτά τα δύο δεδομένα, η αρμοδιότητα συντονισμού που δίνει στην Ένωση η συνθήκη για την οικονομική πολιτική αποκτά πιο δεσμευτικό χαρακτήρα κάπως, με κάποιο τρόπο. Σε μια τέτοια περίπτωση είναι σαφές ότι η απουσία συγκεκριμένου και δέοντος ρόλου του Κοινοβουλίου, στον κοινοβουλευτικό έλεγχο των δράσεων αυτών, που ξεπερνά αυτό που υπήρχε στο προηγούμενο, σε προηγούμενο πλαίσιο μετά το 2010 γίνεται κρίσιμο για την νομοποίηση του Κοινοβουλίου δημοκρατικά. Άρα υπάρχει ένα δημοκρατικό έλλειμμα που πρέπει να καλυφθεί και που μπορεί να καλυφθεί με δύο τρόπους. Αφενός με την αύξηση του ρόλου του Κοινοβουλίου ως decision making, νέες νομικές βάσεις, διαφορετική ερμηνεία από τη φυστάμενη μεταρρύθμιση των ε, συνδικών δύο οργανικές ε, συμφωνίες ή μια άλλη διάσταση που πρέπει την έκθεση Ράγκελ και που δεν καλύπτεται παρκώς τώρα και που αφορά την ερμηνεία της εφαρμογής της έννοιας του πολιτικού ελέγχου και της λογοδοσίας της Επιτροπής ενώπιον του Κοινοβουλίου. Έννοια που φοβάμαι ότι εμφανίζεται εναλλακτικά με την ενίσχυση του ρόλου του Κοινοβουλίου και στα κείμενα της λεγόμενης διαδικασίας Βαν Ρομπάι για την ΟΝΕ. Την ιδέα δηλαδή ότι και σε περιπτώσεις μεταγενέστερης ενίσχυσης του δεσμευτικού χαρακτήρα του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών μέσω αυτών των ε, contract arrangements, ο ρόλος ε, του Κοινοβουλίου, η αύξηση του ρόλου του Κοινοβουλίου μπορεί να περιοριστεί στο γεγονό ότι θα έρχεται η Επιτροπή να λογοδοτεί ενώπιον του Κοινοβουλίου. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, αυτό δεν είναι λύση, αλλά αν συμβεί κάτι τέτοιο είναι σαφές πως η έννοια του πολιτικού ελέγχου και του accountability ε, θα πρέπει να αποτύχει ισχυρότερη παρουσία από την απλή στη χρονική στιγμή της, επιλογής της, επιτροπ... της εκλογής της Επιτροπής. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει στο πλαίσιο αυτό να ενισχύσει και να δώσει στοιχεία που θα δίνουν ουσία στην αυξανόμενη αρμοδιότητα της ε, Επιτροπής στην υλοποίηση στόχων που ξεπερνά αυτούς που αρχικά είχε θέση η Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστούμε. Δεν έχουμε άλλες παρεμβάσεις. Ο κύριος Ζανζέλ για να απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στα βασικά σχόλια του κάθε ομιλητή. Αλλά θα προσπαθήσω και ταυτόχρονα να είμαι πολύ σύντομος. Ξεκινάω από τον κύριο Γκερέρο. Δύο σημεία. Πρώτον, δεν έχει και πολύ δίκιο ο κύριο Γκέρερ, λοιπόν, που το λέω όταν λέω ότι το πρόβλημα με το εκτελεστικό σώμα και την αυτονομία του μοιάζει με τη δημοκρατία της Βαϊμάρης και τα προβλήματα εκεί, ε, λυπούμε, αλλά σφάλει ο κύριος Γκερέρο. Δεν θέλω να γυρίσουμε πάλι πίσω στο 18ο αιώνα, γιατί συνέχεια γι' αυτό τον αιώνα αναφέρομαι, αλλά ένα κοινοβούλιο σαν το δικό μας που αναπτύσσεται, που αναλαμβάνει νέες δυνάμεις, μοιάζει πολύ περισσότερο με τις Βρετανικές εξελίξεις, ε, τις πολιτικές και με τη Γαλλική Επανάσταση ακόμη. Για παράδειγμα, στο Γαλλικό Σύνταγμα. Μετά την περίοδο της τρομοκρατίας, ε, στα τέλη του 17ου, η ανακοινώσεις γίνονταν γραπτός. Δεν επιτρεπόντουσαν προσωπικές ε, επαφές. Κάπως ακραία λύση ήταν αυτή. Μιλώ για τους ε, εκπροσώπους των διαφόρων εξουσιών. Έτσι, λίγο ακραία η διάκριση των εξουσιών σε αυτή την περίπτωση. Ο κύριος Γκερέρο πάλι είπε ότι διαφωνεί μαζί μου σε ένα σημείο που όμως νομίζω ότι συμφωνούμε τελικά, ότι δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ασκεί τον ρόλο που έχει ε, να ελέγχει, ο οποίος θα πρέπει να είναι όμως ενισχυμένος και διευρυμένος. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν, να καλούμε τον πρόεδρο της Κομισιόν να ανακοινώνει το πολιτικό του πρόγραμμα πριν οριστεί. Ε, καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τηρεί κάποιου όρου και προποθέσει. Όλα αυτά τα προβλέπουν οι συνθήκε. Αλλά εγώ τι ήθελα να πω. Ήθελα να πω ότι από τη μία να είναι ένα είδος εκτελεστικού το κοινοβούλιο, ούτε στόχος μου είναι, ούτε στην έκθεση περιλαμβάνεται. Και τον ωφετήχ της Επιτροπής ΑΦΚΟ για τις προτάσεις μομφής κατά επιτρόπων, ούτε αυτό το περιλαμβάνει η έκθεσή μου, για λόγους τους οποίους θα εξηγήσω στον κύριο Νταφ. Πολύ σωστά μας είπε ο κύριος Νταφ, ότι καλύτερα είναι να γίνονται περισσότερες προτάσεις, να διατυπώνονται ιδέες, πιο έτσι ρητές ιδέες, ε, για να τις χρησιμοποιήσουμε στην επόμενη ε, συντακτική συνέλευση. Αλλά εγώ νομίζω ότι μπορούμε ε, να έχουμε υπόψη μας πολλές διαφορετικές δυνατότητες δράσης. Αλλά αν σε μία έκθεση αναφέρουμε το τι θα περιλαμβάνουν οι μελλοντικές συμφωνίες, πάμε σε λάθος κατεύθυνση. Έχουμε τη συνθήκη της Λισαβόνας και πάνω σε αυτήν πρέπει να δουλέψουμε. πάρα πολλές υποδείξεις ή αναφορές σε μια μελλοντική συμφωνία θα αποδυνάμωναν κατ' εμέ την έκθεση, διότι κάτι τέτοιο θα σήμαινε ότι τα άλλα θεσμικά όργανα, Συμβούλια και Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας υποχρέωναν να διεξάγουμε εργασίες, εκθέσεις για την επόμενη ε, συντακτική συνέλευση αλλά πρέπει να είμαστε και μετριοπαθείς και συγκρατημένοι. Πρέπει να επιδείξουμε αυτοσυγκράτηση σε ό,τι αφορά τι μελλοντικέ συμφωνίε και συντακτικέ συνελεύσει. Και σε σχέση με κάτι που είπε ο κύριο ε, Σέφλιν, ότι πρέπει να εκπροσωπούμε τα δικά μας ε, κοινοβούλια και όχι αυτά τα οποία θα συγκληθούν μετά ή θα συγκροτηθούν μετά τι εκλογέ. όπως και στην περίπτωση ε, της κληρονομιάς ε, που πρέπει να τη δεχθεί η μη ο κληρονόμος ε, θα μπορούσε το επόμενο κοινοβούλιο να μην δεχθεί αυτά που θα του κληροδοτήσουμε άρα να μην καταλήξουμε σε ακραίες λεπτομέρειες Τώρα για τους νεοεκλεγέντες. Μα όλοι είναι νεοεκλεγέντες κύριε Γκουαλτιέρη. Όσοι έρχονται ξανά ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει σημασία το αν ήταν βουλευτές από το 79 ή αν ήταν 2, 3, 4 θητείες. Ήρθαν ξανά στο Κοινοβούλιο γιατί τους ξαναψήφισε το εκλογικό σώμα και τους έδωσε εντολή να εκπροσωπήσουν ε, αυτούς τους πολίτες. Άρα είναι νεοεκλεγέντες. Παρόλα αυτά έτσι ερχόμαστε όλοι στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο ως νεοεκλεγέντες. Τώρα, η αγγλική εμπειρία τι μας έχει δείξει. Το τέλος αυτής της όλης διαδικασίας με τις προτάσεις ε, Μομφής και όχι το αντίθετο. Σας δίνω ένα παράδειγμα τη μείωση του μισθού ενός ε, υπουργού. Ακούστηκαν πολλά και διάφορα, δεν με εκπλήσουν βέβαια, αλλά το ότι τελικά δεν πιστεύουν οι ίδιοι βουλευτές ε, την πολιτική τους ιδιότητα. Δεν έχουν εμπιστοσύνη και πρέπει να αποταθούν στα εθνικά κοινοβούλια. Ή ότι μπορεί ένα, δύο, τρία κόμματα να ζητήσουν παρέτηση ενός υπουργού. Δεν σημαίνει ότι θα το κάνει αυτό ο υπουργό, αλλά σίγουρα έχει μεγάλο βάρος ε, μετά. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε και εμείς ότι αν η ε, Κομισιόν ε, ή κάποιος επίτροπος δεν πηγαίνει καλά, δεν τα κάνει σωστά, να πάμε στην Κομισιόν και να πούμε ότι θα πρέπει ίσως αυτός ο επίτροπος να ε, αποχωρήσει, να παρετηθεί. Εγώ μπορώ αύριο να πάω στους δημοσιογράφους και να καταγγείλω οποιονδήποτε, τον πρώτη Κομισιόν, να ασκήσω κριτική. Δεν θα επηρεάσει τίποτα αυτό. Γιατί δεν υπάρχει κάποια επίσημη διαδικασία που θα μπορούσε να ακολουθηθεί γι' αυτό και λέω ότι είναι σημαντικό ο πρόεδρος της Κομισιόν να είναι αυτόνομος, να έχει αυτονομία. Έχει μένα, αλλά είναι πάρα πολύ περιορισμένη. Ο κύριος Χέφνερ νομίζω το είπε πολύ ξεκάθαρα, ότι αυτή τη στιγμή μας ανησυχεί ότι μη μπορεί η Επίτροπη οι επίτροποι να ορίζονται από τα κράτη-μέλη και τελικά να τους επιβάλλουν στον πρώτη της Κομισιόν αυτούς τους επιτρόπους. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να έχει ελευθερία επιλογής ο πρόεδρος, να διαλέγει τους δικούς του επιτρόπους. Και νομίζω αυτό είπε και ο κύριος Μπροκ. Κάτι ενδιαφέρον που έχω παρατηρήσει είναι ότι οι Γερμανοί συνάδελφοι, παρά το γεγονό ότι μπορεί να από διαφορετικό πολιτικό υπόβαθρο, είναι όλοι, μάλλον όχι αντίθετοι, τέλο πάντων έχουν επιφυλάξεις ε, στην, απέναντι στην ιδέα των επιτρόπων άνευ χαρτοφυλακίου και κατά της ε, εναλλαγής των επιτρόπων. Σαν να μην είναι κάτι φυσιολογικό αυτό το σύστημα. Λες να μην υπάρχει στην Πολωνία, στη Γαλλία, στην Ισπανία ή σε άλλες χώρες το να μην έχουν ποτέ επίτροπο οι χώρες αυτές ε, θα ήταν ε, για αυτές κάτι πάρα πολύ αρνητικό. Ούτε θέλουμε να έχουμε χώρες πρώτης κατηγορίας, δεν χώρες δεύτερης κατηγορίας. Ε, θέλω λοιπόν να πω το εξής, πάρα πολύ ξεκάθαρα. Εγώ δεν είμαι υπέρμαχος της ιδέας ή τέλο πάντων άκρο ενθουσιώδη απέναντι στην ιδέα αυτή τη αναλλαγή επιτρόπων ή των επιτρόπων, μάλλον άνευ χαρτοφυλακίου. Απλά λέω ότι είναι μια ιδέα πρακτική, η οποία θα επιτελέσει δύο λειτουργίε. Η πρώτη θα εξασφαλίσει τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του έργου της Επιτροπής και δεύτερη θα εξασφαλίσει ότι όλες οι χώρες θα έχουν έναν επίτροπο. Είναι κάτι που έχει ζητηθεί. Ρητό μάλιστα με το Ιρλανδικό δημοψήφισμα. Και κανεί δεν ήταν ικανοποιημένο με τη λύση τη Λισαβόνα που μείωνε τον αριθμό των επιτρόπων. Ο κ. Σχέφνερ λέει ότι θα είναι πολύ περίεργο. Μα υπάρχουν χιλιάδε παραδείγματα υπουργών άνευ χαρτοφυλακίου στις εθνικές κυβερνήσεις. Μπορεί να μην είναι 7 ή 8, εν γέννη είναι 1 ή 2, ανάλογα με τη χώρα, αλλά υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, υπάρχουν πάρα πολλοί υπουργοί άνευ χαρτοφυλακίου. Μπορεί να μην λέγονται έτσι, να μην του αποκαλούν έτσι σε κάποιες περιπτώσεις. Να είναι ένα είδος υφυπουργού. Τι κάνει, ας πούμε, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Δεν έχει καθορισμένο ρόλο. Και άλλα παραδείγματα έχουμε εκτελεστικούς φορείς, εκτελεστικά σώματα, όπου υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν κάποια συγκεκριμένη αρμοδιότητα, έχουν σκιώδεις δε ε, υπουργού στην αντιπολίτευση. Ο ρόλος του εκτελεστικού δεν ορίζεται μεν επαρκώς ξεκάθαρα, αλλά υπάρχει και μπορούν να κάνουν κάποια πράγματα. Μπορούν να εκπροσωπούν την Κομισιόν. Οι Επίτροποι Ανευχαρτοφυλακίου μπορούν να εκπροσωπούν την Κομισιόν σε εξωτερικό ή και εντός της Ένωσης, όσο οι άλλοι επίτροποι χειρίζονται τα χαρτοφυλακιά τους. Και επομένως οι επίτροποι αν δεν θα μελετούν τους δικούς τους φακέλους αφού δεν έχουν χαρτοφυλάκιο, αλλά τα σημαντικότερα θέματα των άλλων επιτρόπων. Τα βασικά ζητήματα δηλαδή που απασχολούν την Κομισιόν. δεν τη θεωρώ τόσο πολύ είτε τολμηρή, είτε ρηψοκίνδυνη, είτε παράδοξη αυτή τη λύση. Τη θεωρώ απλά μια λύση. Η καλύτερη ίσως προσέγγιση θα ήταν να μείνουμε στο πνεύμα και το γράμμα της συνέντευξης Λισαβόνας. Τότε όμως τι θα συνέβαινε, σε κάποια χρόνια, 6-7 χώρες δεν θα είχαν επίτροπο και αυτό ξέρουμε ότι δεν είναι επιτρεπτό λόγω των πολιτικών ευαισθησιών. Με τη λύση που προτείνω λοιπόν δεν θα στερήσουμε επιτρόπους από τις χώρες, αλλά θα βελτιώσουμε και την αποτελεσματικότητα της Κομισιόν. Απλά κάποιοι θα είναι άνευ χαρτοφυλακίου. Τώρα να κάνω κάποια σχόλια ως προς τον κύριο Λάινεν να του θέσω υπόψη το εξή. Ίσως να μην έχει παρακολουθήσει ακριβώς το ρυθμό της έκθεσης και να μην έχει αντιληφθεί τι κρύφθηκε πίσω από τους υποτίτλους που δώσαμε στην έκθεση. Αυτό έγινε συνδρίες των συντονιστών συγκεκριμένα, όπου δόθηκε πολύ αυστηρή εντολή να συζητηθούν οι σχέσεις του Κοινοβουλίου με την Κομισιόν και τίποτε παραπάνω. Φυσικά και υπάρχει ένα εκατομμύριο άλλα πράγματα που θα ήθελα εγώ να συζητήσουμε πέραν αυτό. Αλλά αφού αυτή τη δέσμευση ανέλαβα, έτσι πρέπει και να κάνω. Ναι, μεν ο τίτλος είναι ευρύς, οι υπότιτλοι, οι είναι πιο περιορισμένε φυσικά. Οι σχέσεις μεταξύ Κοινοβουλίου και Κομισιών έχουν αποτελέσει αντικείμενο εκατοντάδων χιλιάδων λέξεων, διατριβών ε, ε, σε όλο τον κόσμο. Δεν ξέρω, μπορεί ο κύριος Λάινεν να θεωρεί δεν διάβασα την έκθεσή του. Αν τη διάβασα, τη διάβασα και πάρα πολύ προσεκτικά μάλιστα. Το θέμα είναι τι προσέγγιση πρέπει να ακολουθήσουμε τώρα. Από εδώ και πέρα. Νομίζω αν θέλουμε μια πιο τεχνοκρατική, νομικήστικη κομισιόν ή αν έχουμε μια έκθεση που απλά θα αναφέρει τι, εκθέσει, τι βελτιώσεις και διαφορές ε, έχουν ε, προκύψει μετά την συνθήκη της τα κτλ. Θα τα μια δυνατότητα, αλλά εμείς θέλουμε να εστιάσουμε στα βασικά συνταγματικά ζητήματα. Κατά πρώτο και κύριο λόγο, διότι όλα τα άλλα μπορούν να είναι και αντικείμενο διαπραγμάτευση. Ο τρόπο με τον οποίο τα μεγάλα αυτά προβλήματα τα αντιμετωπίζονται είναι πιο σημαντικό από το να δούμε μετά τι τεχνικέ λεπτομέρειε. Είμαι ευγνώμων στον κύριο Σέπφλιν για την ιδέα. Το θέμα της συγκυρίας που ανέφερε είναι σημαντικό. Στο Κοινοβούλιο πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν ένα κοινοβούλιο κλείνει τη θητεία του έχει άλλη οπτική από ότι ένα επερχόμενο κοινοβούλιο. Γι' αυτό, ακριβώς γι' αυτό, ο κύριος στόχος μας στους επόμενους μήνες είναι να επικεντρωθούμε στα ζητήματα ορισμού Πρόεδρου της Επιτροπής, ορισμού Επιτρόπων, Framework Agreement, παρουσίαση καθοδηγητήριων γραμμών. Αυτό είναι φυσικό βέβαια. Γιατί αυτό που θέλουμε να δημιουργήσουμε είναι ένα είδος θεσμικής νομολογίας για τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί η συνθήκη της Λισαβόνας στον ορισμό της πρώτης νέας επιτροπής μετά τη συνθήκη. Γι' αυτό υιοθετήσαμε την προσέγγιση αυτή. Αυτή ήταν η προοπτική που είχα, γιατί εκεί θεωρώ ότι πρέπει να επικεντρώσουμε. Το Κοινοβούλιο θα μπορεί ενδεχομένως να διαμορφώσει μία νομολογία και να αφήσει αυτό ως ε, κληρονομιά για το μέλλον. Και αυτό το θεωρώ σημαντικό για μένα. Κοιτάξτε, ε, έχω να κάνω και άλλη δουλειά, δηλαδή πρέπει να κάνω αναγγελίες. Μπορείτε να τελειώνετε λοιπόν. Έλεγα ότι ακούστηκαν πολλές προτάσεις Γουαντιέρι, Brock, που πρέπει να τις εξετάσουμε πιο διεξοδικά. Κλείνω. Νομίζω απάντησε σε όλους. Πιστεύω ότι τώρα μπορούμε να συζητήσουμε βάση της έκθεσης. Προσπάθησα να σας εξηγήσω γιατί έκανα τις επιλογές αυτές. Δεν ήταν επιλογές που έγιναν τυχαία ή ελαφρά την καρδία. Ευχαριστώ όλους για τα επικριτικά και θετικά σχόλιά σας. Θα ξεκινήσουμε μια ανοιχτή συζήτηση με τους σκιώδεις ηγητές και τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους για να ακούσουμε τις απόψεις όλων και να βρούμε μια συνένεση που θα επιτρέψει να δημιουργήσουμε τους επόμενους μήνες μια βάση μελλοντικών εργασιών. Ευχαριστώ για την πληρέστατη παρουσίασή σας. Πρέπει να θέσουμε προθεσμίες. 23 Ιανουαρίου του 2014 προθεσμία για τις τροπολογίες. Κοντά είναι η προθεσμία, αλλά μόνο έτσι μπορούμε να ψηφίσουμε σε αυτή τη θητεία. Το Φεβρουάριο ψηφίζουμε. Προτείνω να κάνουμε μία ακρόαση για αν χρειαστεί μέσα στον Ιανουάριο. Να σας ενημερώσω επίσης για τη συνάντηση των συντονιστών για να υπάρξει επικύρωση της απόφασης των αποφάσεων από, τους, ε, από την ε, Επιτροπή. Ορίστηκαν μια σειρά εκθέσεων. ΕΛΚ, ο υποφαινόμενος, αναλαμβάνει την έκθεση για την πρωτοβουλία για τη σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκού και Εθνικών Κοινοβουλίων. Για το θέμα της έδρας, η πλειοψηφία των συντονιστών δεν θέλησαν να υπάρξει μια έκθεση πρωτοβουλίας για την αλλαγή των συνδικών σχετικά με την ενιαία έδρα. Επίσης προτείνουν να ανατεθεί η έκθεση για το άρθρο 127 του κανονισμού την αλλαγή των ε, διοργανικών συμφωνιών ε, και την καταγραφή του στο Μητρό Αδιαφάνεια στην ομάδα των σοσιαλιστών με εισηγητή τον κύριο Γκουαλτιέρη. Για τις αλλαγές που είναι αναγκαίες στον κανονισμό για να εισαχθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής υπογραφής δεν υπάρχει ακόμα το όνομα του εισηγητή αλλά προτείνεται να δοθεί στο ΕΛΚ η έκθεση. Η πρόταση να ανατεθεί έκθεση στον συνάδελφο Σόλτς της ΓΚΟΕ για την γνωμοδότηση πρωτοβουλίας της Οικονομικής Επιτροπής για τον ρόλο της Τρόικας. Προτείνεται να δοθεί σε αυτούς. Για το πρόγραμμα της ε, ζώνης ευρώ και της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης ζώνη ευρώ είναι ο κύριος Νταφ. Κατόπιν έκθεση για την Επιτροπή Προπολογισμών για τις διαπραγματεύσεις του πολιετού οικονομικού προγράμματος 2014-20 και τις προοπτικές. Τώρα, έκθεση άρθρου 2.11 παράγραφος 7 για τον κανονισμό αποφασίσει και να περιμένουμε την επιστολή του Προέδρου που θα έπρεπε να αναφέρει καλύτερα το περιεχόμενο της έκθεσης που να σας πω την αλήθεια ήταν αρμοδιότητα του Προέδρου, σε μένα είχε ανατεθεί, αλλά υποφάσισα να αναβάλω την εξέταση. Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία. Ο Χέφνερ θα παρακολουθεί τις διαδικασίες και θα ενημερώνει τις αρμόδιες ε, δομές και την Επιτροπή μας για τις προτάσεις για την ακρόαση. Ο κ. Χέφνερ ανέλαβε την ευθύνη της πρωτοβουλίας αυτής. Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της συνθήκης της ε, Λισαβόνας, είπαμε ακρόαση 20 Ιανουαρίου, υπάρχει συμφωνία με το πρόγραμμα που προτείνει ο εισηγητής. Σε ό,τι αφορά το μέλλον της, Ευρώπης, άλλη ακρόαση που θα γίνει το Μάρτιο, η έμφαση θα, στις θα είναι η πρόταση τροποποίησης εθήκης που που δημοσίευσε η Επιτροπή, που κυκλοφόρησε η Επιτροπή, με υπόσχεση παρέμβασης και του Προέδρου Μπαρόζο, οπότε θα κληθεί ο κύριος Μπαρόζο. Πάντως υπάρχει, θεωρείται ότι θα υπάρξει πρόταση της Επιτροπής από πλευράς ε, του Αντιπροέδρου ή του Προέδρου δεν θα επιτρέψουμε να προχωρήσει η ακρόαση ενός Έλληνα πολίτη που ζητούσε να υπάρξει ένα παγκόσμιο φιλοσοφικό συνέδριο. Θα την περάσουμε στην Επιτροπή Αναφορών. Να σας πω επίσης ότι υπάρχει ένα κείμενο του κυρίου Σκοτσέζε ενός, συγγνώμη, ενός σκότου πολίτη που αφορά ε, την εξέλιξη, την κατάσταση της σκοτίας σε περίπτωση ε, απόσχησής της από τη Μεγάλη Βρετανία. Αυτό θα το αναβάλαμε για μετά. Να μιλήσουμε τώρα για την διευθυντική έκθεση σχετικά με το ρόλο και τις δραστηριότητες της Τρόικας όσον αφορά τις χώρες του προγράμματος της Ευρωζώνης. Λείπει όμως ο εισηγητής Είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν να αναβάλουμε την έκθεση αυτή για την επόμενη συνάντηση. Αλλά έχω το χρόνο να σε ευχηθώ καλά Χριστούγεννα, ευτυχές το νέο έτος, ό,τι καλύτερο μπορείτε και έχετε τη δυνατότητα για τις διακοπές σας. Καλά Χριστούγεννα.